Ja, Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε σας παρακαλώ, να έχουμε λίγη τάξη στην αίθουσα, να επανέλθουμε. Έχω μια καλή είδεση. Κύριε Ριβελίνη, για σας σας ενδιαφέρει. Η ημερομηνία για την ψηφοφορία για τις δύο σας εκθέσεις έχει πλέον καθοριστεί. 26 Σεπτεμβρίου το βράδυ στις 7 η ώρα στο Στρασβούργο. Μια μεγάλη αίθουσα 20 γλώσσες, διερμηνές σε 20 γλώσσες. Θα ψηφίσουμε λοιπόν στις 26 Σεπτεμβρίου τη Δευτέρα του Στρασβούργου στην αίθουσά σας. Σας παρακαλώ καταγράψτε το. Okay. Χαμπέμους Πάπα, λέει ο κύριος Ζιβελίνη. Χαμπέμους Πάπα. Χαμπίους Πάπα, Έχετε, έχετε Πάπα. Βγήκε άσπρος καπνός, λέει ο κυριο Σέστας. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη, στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Τώρα είναι η δική μου γνωμοδότηση η οποία πρέπει να ψηφιστεί για τις, για τις δημόσιες προμήθειες. Νομίζω ότι έχετε ένα κατάλογο Έχετε τον κατάλογο ψηφοφορίας. Έχω κοιτάξει τις τροπολογίες. Ελπίζω ότι σας ικανοποιούν οι προτάσεις μου. Δεν είμαι πολύ καλά ικανοποιημένος με το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 6 και έχω κάποιες ερωτήσεις για την τροπολογία 20 του κ. Κονσουλίνο, Κοτσολίνο. Εδώ ήταν ο κ. Κοτσολίνο, αλλά φαίνεται ότι έχει μόλις φύγει. Πάντως έχουμε συζητήσει για το θέμα αυτό. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν <clears throat> σχόλια μπορούμε να ξεκινήσουμε ψηφοφορία. Όχι, εντάξει, ξεκινάμε. Είναι η δική μου έκθεση λοιπόν όπως σας είπα, τροπολογία 1. Σας παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια. Αν είναι σαφή τα πράγματα δεν χρειαζόμαστε ψηφοφορία ηλεκτρονική. Τροπολογία 1, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Παράγραφος 1α, τροπολογία 2. Στας ή τελαζ Μπαλτσίτης ψηφιπέρ κατά αποχές δεκτή. Παραγραφος 2 τροπολογίες 3 και 4 που είναι συμβατές. Ιβανόβα και Μακοβέη ψηφιπέρ κατά αποχές δεκτές. Τροπολογία 5 και 6 που είναι ταυτόσιμες αλλά χρειάζεται χωριστή ψηφοφορία εδώ κατά τμήματα. Την 3 και την 4 τις έχουμε ψηφίσει και εγκρίθηκαν. Θέλετε χωριστή ψηφοφορία. 3 και 4 έχετε υπερψηφίσει, εντάξει. 5 και 6 τώρα είναι ταυτόσιμες, αλλά υπάρχει χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα των 5 και 6. Considers μέχρι corruption. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θέλουμε ηλεκτρονική επαλέθευση. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όχι, όχι, δεν μπορώ να πω ποιος είναι κατά για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κλείνω την ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα. Μπορούμε να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 5 και 6 καλεί την Κομισιόν μέχρι διαδικασίες ψήφι υπέρ κατά απόχες και αυτό το τμήμα απορρίπτεται τροπολογία 7 στην παράγραφο 2α Μπαλτσίτης υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται 8 Μακκοβέι υπέρ κατά αποχές και αυτή η Τροπολογία 9 και 10 είναι ταυτόσιμες στην παράγραφο 4. Πάξας και Ιμπράσας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας ψηφοφορίες. Το αποτέλεσμα είναι ότι εγκρίνονται 13-9. <clears throat> Τροπολογία 11, Μακοβέη, μια νέα παράγραφος, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12, Φιέλνερ, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13. Κοτσολίνο, ψήφι Κατά. Απόχες, απορρίπτεται. 14, Αγιάλα Σέντερ, υπέρ. Κατά. Απόχες και αυτή απορρίπτεται παραφο 5 5α, νέα, τροπολογία 15, Ιβάνοβα. Θέλετε έλεγχο για τη 14, βεβαίω. Θα κάνουμε έλεγχο στην τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Νομίζω ότι η Φιλελεύθερη και το ΕΛΚ είχαν την πλειοψηφία, μπορεί και όχι. Άρχεται η ψηφοφορία, απορρίπτεται λοιπόν. Απορρίπτεται παρόλα αυτά. Είχατε δίκιο να ζητήσετε έλεγχο. Τροπολογία 15 Ιβάνοβα. Μια 5, παράγραφος 5α υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 16 Μπαλτσίτης υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 17 Πολωνομάδων ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18, πάλι μια κοινή τροπολογία, στάση, τα λαμπατζίτς κτλ. Υπέρ, κα, υπέρ, υπέρ, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 19 εκπίπτει λόγω της έγκρισης 18. Πάμε τώρα στην τροπολογία 20, δεύτερο τμήμα. Κότσολίνο. Το πρώτο τμήμα εκπίπτει μετά την έγκριση της 3. Ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογία, το οποίο μας δεν ψηφίζεται, και το τρίτο τμήμα, ε, το οποίο εκπίπτει, το οποίο μάλλον ψηφίζεται σαν ε, προσθήκη 18. Κατά αποχές χρειαζόμαστε ηλεκτρονικό έλεγχο. Τρίτο τμήμα της τροπολογία 20 Κοτσολίνο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21, Σέντεργαρτ. ψηφιπέρ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική. Διαδικασία άρχεται η ψηφοφορία. 23 έχουν λάβει μέρος στη ψηφοφορία ομόφωνα υπέρ. Σας ευχαριστώ λοιπόν και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σημείο 6 τώρα. Πάλι έκθεση Bad συνεγνωμοδότηση για το ΦΠΑ. Έχουμε λοιπόν μία σειρά τροπολογίες Θέλετε να ψηφίσουμε από κοινού. Όχι, θα ψηφίσουμε τώρα. Παράγραφό 1, τροπολογία 1, μπαλτσίτη. Υπέρ. Κατά. απόχε. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά πρέπει να το ξανακοιτάξουμε. Ηλεκτρονικό έλεγχο Άρχεται η ψηφοφορια περα Πέρας. 12-10 εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Η ένα έχει δεκτή. Τροπολογία 2. μπράσα Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Πάξα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Φιλελεύθερη και έλεγχη είναι κατά, αλλά χρειαζόμαστε ηλεκτρονικό έλεγχο. Τροπολογία 3 με ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται. Κυρία Χολμάιερ, έχετε ψηφίσει κατά. <clears throat> Κλείνω την ψηφοφορία. Α, ψηφίσει η κυρία Χολμάιερ με την κάρτα της. 24 ψήφισαν, 11, 13 απορρίπτεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 4. 4 και 5 ψηφίζουμε χωριστά 4 ψήφι υπέρ. 4. Παλτσίτες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 ημπράσας υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 Μπαλτσίτης υπέρ κατά εγκρίνεται. Παράγραφος 4 τροπολογία 9 9, 7 και 8 μπορούν να, να συνδυαστούν, αλλά θέλετε να ψηφίσουμε χωριστά. Εντάξει, 9. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Μπαλτσίτης υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Ιμπράσες υπέρ. Κατά. Αποχές πρέπει να δούμε με ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 8. 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απέριπτε. Παράφωση 6 τροπολογία 10. Ήμπρασας. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 που μπορεί να συνδυαστεί με τις άλλες τροπολογίες. Ψηφίζουμε χωριστά. 11 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 12. Αγιά Σέντερ υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Θέλουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 12 Αγιά Σέντερ. Λοιπόν, τροπολογία 12, ηλεκτρονικός έλεγχος, πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Παράγραφος 6, τροπολογία 13, Ιάν Μιλντερ, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 7, τροπολογία 14, Πάξας, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 8, τροπολογία 15, Μπαλτσίτης, υπέρ. Κατά. Αποχές γίνεται δεκτή. Παράγραφος 10, τροπολογία 16, συμβράσες. υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17, Μπαλτσίτης, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 18 τσεσκοβα υπερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράφος 10α, τροπολογία 19, Τσεσκόβα. Υπέρ, κατά, απόχε, Είναι πολλέ οι αποχέ, δεν ξέρω τι ακριβώ είναι. Πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. 19 Τσέσκοβα. 19 Τσέσκοβα. Ηλεκτρονικό έλεγχο. Πέρα. Απολύτω. Παράγραφο 20 του εισηγητή ψήφι περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και εδώ ομοφωνία. Ωραία. Το επόμενο σημείο της μέσης διάταξης. Καταρχήν συγχαίρω τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο σημείο της Μέσης διάταξης είναι το σημείο 7. Είναι η μελέτη που έχουμε ζητήσει να συνταχθεί από την Blomeyer και Sands για την ε, προενταξιακή χρηματοδότηση για την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Έχουμε μαζί μας ως προσκεκλημένο τον κύριο Άκερμαν, ο οποίος θα μας κάνει μια παρουσίαση ισχυρού σημείου και θα παρουσιάσει την έκθεση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αυτή η μελέτη έγινε μεταξύ του Δεκεμβρίου 2010 και του Μαρτίου του 2011 και η έκθεση παρουσιάστηκε το Μάρτιο. Η παρουσίαση έχει τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα μιλάει για τους στόχους και την μέθοδο που είναι σύντομο. Το, τα άλλα δύο τμήματα για τα πορίσματα και τα διδάγματα είναι λίγο πιο μακροσκελή. Η στόχη, λοιπόν, καταρχάς, ήταν να καταλάβουμε αν η εμπειρία από την πρωταξιακή διαδικασία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες χώρες και σε ποιο βαθμό αυτή η εμπειρία έχει όντως ε, εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες. Και για να ε, απαντήσουμε, εστιάσαμε στα μαθήματα και στα διδάγματα που αφορούν δύο θέματα τη διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και την συνεισφορά αυτών των κονδυλίων προενταξιακής βοήθειας στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία για να δημιουργήσει δομές που, όπως προβλέπουν τα διαφθορτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Η μέθοδος. Εφαρμόσαμε μια κλασική συνηθισμένη μέθοδο με μια έρευνα γραφείου ε, επιτεκμηρίωσης που αφορά τις ε, χώρες που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και το 2007. Έγινε μια έρευνα ε, online από εκπροσώπους των υποψηφίων χωρών και δυνητικά υποψηφίων χωρών και είχαμε άμεσες διαβουλεύσεις με 23 ενδιαφερομένους φορείς από τη Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Ισλανδία και τις υπηρεσίες κομισιών και δύο μελέτες περιπτώσεων για την Κροατία και την Ισλανδία. Να περάσω στα πορίσματα τώρα. Αυτά τα ιστογράμματα σας, δίνουν, δείχνουν τη συνολική χρηματοδότηση ε, προενταξιακά ε, από το 2003 μέχρι το 2007 στην Ρουμανία και Βουλγαρία. Ε, δεξιά τα κίτρινα ιστογράμματα σας δείχνουν κάθε χρόνο πόσα δόθηκαν και τα πράσινα αριστερά τα πραγματικά ποσά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Συνολικά η Ρουμανία πήρε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή την περίοδο. Περίπου το 95% χρησιμοποιήθηκε, με Βουλγαρία πήρε περίπου α, μισό δις ευρώ και το 86% περίπου χρησιμοποιήθηκε. Να, αν δούμε την απορρόφηση ετήσια βάση, η Ρουμανία είχε μια σταθερή πορεία από το 2003 μέχρι το 2007, ενώ η Βουλγαρία δεν ήταν τόσο σταθερή, είχε μεγάλη πτώση στην απορρόφηση το 2006, ε, όπου το 60% των κονδυλίων μόνο απορροφήθηκαν. Συγκρίναμε επίσης το ποσοστό ε, απορρόφησης με την κατάσταση των χωρών που εντάχθηκαν το 2004. Και ε, κάνουμε μια χαρτογράφηση σε σχέση με τη χρονιά ένταξης και είδαμε τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια τι ακριβώς συνέβη πριν την ένταξη δηλαδή. Οι επιδόσεις της ε, Ρουμανίας είναι αντίστοιχες με των χωρών που εντάχθηκαν το 2004 με μια ελαφρά αύξηση τη χρονιά τη ένταξη σε σχέση με τι χώρε που εντάχθηκαν το 2004. Ενώ η Βουλγαρία βλέπουμε ότι οι επιδόσεις ήταν πάλι ασταθεί κάτω από τη μέση επίδοση των χωρών που εντάχθηκαν το 2004 και όπως ανέφερα και προηγουμένως, μία χρονιά πριν από την ένταξη υπήρχε μία φοβερή μείωση, σημαντική μείωση στην απορρόφηση. Εντοπίσαμε τώρα διάφορα διαφθορτικά εμπόδια σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πρωταξιακών κονδυλίων. Το πιο σημαντικό είναι η πολιτική φύση της αλλαγής που συνέβη στη δημόσια διοίκηση που δεν είχε γίνει πλήρως κατανοητή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Και ίσως αυτό οδήγησε σε μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το τι μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα πολύ μικροφωνικό διάστημα. Δεν έλαβαν επαρκώς υπόψη τη διαδικασία αλλαγής του τρόπου διαχείρισης, του τρόπου διοίκησης. Και δόθηκε μεγάλη έμφαση στην εκταμείευση και όχι στις επιπτώσεις. Αυτό αφορά όχι μόνο τις υποψήφιες χώρες, αλλά τις υπηρεσίες της Κομισιόν και τις αντιπροσωπείες της Κομισιόν. Ε, και αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει, δεδομένου ότι όλοι όσοι ενεπλάξαν ε, λειτουργούσαν υποπίεση, τεράστια πίεση, να, για να εκταμιευθούν αυτά τα προενταξιακά κονδύλια. Οι δομές οι οποίες δημιουργήθηκαν για τη διαχείριση των κονδυλίων αυτών προενταξιακής βοήθειας ε, δεν είχαν επαρκείς πόρους και αυτό τελικά μας οδηγούσε σε δουλειά της τελευταίας στιγμής για να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια πριν από την καταληκτική ημερομηνία για να συναφθούν τα κονδύλια κτλ. Και αυτό είχε επίπτωση στο... και στα κονδύλια. Από πλευράς κομισιών εντοπίσαμε απροθυμίες ε, να αφήσουν προγράμματα απλώς να αποτύχουν είχε, υπήρχε υπερβολική εμπλοκή των αντιπροσωπιών ε, στη διαχείριση των ε, των σχεδίων δηλαδή, και αισθανόταν πίεση να μην αφήσουν τα σχέδια αυτά, τα project να αποτύχουν. Υπήρχαν αδυναμίες λοιπόν στο σύστημα και σημαντικά διδάγματα δεν είχαν απορροφηθεί και δεν είχαν, ε, δεν είχαν, δεν είχαν αλλάξει οι συμπεριφορές. Γενικά υπήρχε μια έλλειψη εξέλιξης, αν θέλετε, και από τις υποψήφιες χώρες και από τις ε, υπηρεσίες της Κομισιόν. Δεν άλλασαν συμπεριφορά σε ό,τι αφορά την ε, χρηματοδότηση αυτή. Στις υποψήφιες χώρες οι ενδιαφερόμενοι είπαν ότι τότε αλλά και σήμερα ακόμα υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτικών και των δημοσίων υπαλλήλων που δημιουργεί μια κατάσταση όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι βασίζονται πάρα πολύ σε κανόνες υπερβολικά περίπλοκους για τη διαχείριση των προταξιακών κονδυλίων. Τομεακή παρακολούθηση και η αξιολόγηση. Αυτή ήταν αρκετά αδύναμη γενικά. Επίσης η διαχείριση και οι δομές ας πούμε, ελέγχου και διοίκησης, δεν μιλάω για τους ανθρώπινους πόρους, αλλά για τις δομές, ήταν αδύναμες και ανεπαρκή συχνά για το, τα καθήκοντα. Το βασικό θέμα ίσως αφορά αυτό που είπα στην αρχή, το σημείο αφετηρίας δηλαδή. Όταν ξεκίνησε η προενταξιακή χρηματοδότηση, οι δύο χώρες, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, είχαν κάποια συστήματα τόσο διαφορετικά από αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπήρχε τεράστια πίεση και στις δύο χώρες να κάνουν ε, ταχύτατες αλλαγές για να μπορέσουν να εφαρμόσουν την προενταξιακή χρηματοδότηση με βάση τις ε, ενωσιακές ε, προϋποθέσεις. Οι ανθρώπινοι πόροι. Τεράστιο εμπόδιο στη διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων. Τα βασικά θέματα είναι η χαμηλή μισθή, ε, οι αντικαταστάσεις λόγω από πολιτικούς, γινόταν αρκετά συχνά, παρεμβάσεις πολιτικών και αντικαθιστούσαν τους υπαλλήλους. Γενικά, ε, το επίπεδο management από τους υπαλλήλου ήταν κακό ε, και δεν θεωρείται ότι ήταν σημαντικός ε, παράγοντας. Στη Βουλγαρία ειδικά υπήρχαν τεράστια επίπεδα αποχώρησης των εκπαιδευμένων εργαζομένων με υψηλά προσόντα και δεξιότητας ήδη από την αρχή της δεκαετίας του 90. Πάμε τώρα στη συνεισφορά που είχαν αυτά τα κονδύλια προενταξιακής βοήθειας για τη δημιουργία δομών ε, ανάλογες με αυτές που προβλέπουν τα διαφορετικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Εδώ υπήρχαν διάφορα προβλήματα. Συνολικά η το διοικητικό δυναμικό ήταν ασθενές και αδύνατο να χρησιμοποιήσει, αδύναμο να χρησιμοποιήσει την ε, χρηματοδότηση αυτή με το βέλτιστο τρόπο. Υπήρχαν δυσκολίες στη δημιουργία μηχανισμών συντονισμού ανάμεσα στους διάφορους φορείς που έπρεπε να συνεργαστούν όμως μεταξύ τους. Η οικονομική διαχείριση και οι δομές ελέγχου ήταν ασθενείς, ιδίω η έκθεση των υπηρεσιών της Κομισιόν αναφέρεται συχνά σε δυσκολίες, ιδίως στη Βουλγαρία, για να εντοπίσει και να ε, σταματήσει τις παρατυπίες. Και οι δύο χώρες είχαν προβλήματα να δημιουργήσουν ποιοτικά, να προωθήσουν ποιοτικά σχήματα, project, και προβλήματα με την νομοθεσία για τις προϋποθέσεις των διαρθρωτικών και ταμείων και ταμείων συνοχής, ε, η εδαφική οργάνωση ε, και ο τρόπος ταξινόμησης των ΝΑΤΣ ε, συναντούσε δυσκολίες Επίσης, η δημιουργία τέτοιων ε, δομών διαχείρισης, όπως προβλέπει το ταμείο, ε, συνοχή στο ταμείο, τα διαφορετικά ταμεία, ήταν ε, προβληματική. δεν ξέραμε ποιος είναι υπεύθυνο. Ε, δεν ξέραμε ποιος θα κάνει τις αναφορές, ποιος θα λογοδοτήσει. Και στις δύο χώρες υπήρχαν δυσκολίες να εφαρμοστεί η αρχή της εταιρικής σχέσης, ούτως ώστε όλοι όσοι έπρεπε να εμπλακούν, να εμπλακούν στη διαδικασία προγραμματισμού. Όπως είπα και προηγουμένως, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση ήταν αδύναμη για τη διαχείριση των προεταξιακών κονδυλίων, αλλά οι εκθέσεις της Κομισιόν δείχνουν ε, μικρή πρόοδο για την δημιουργία των απαραίτητων συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγηση, όπως προβλέπουν τα ταμεία. Δεν θα μπω τώρα στον κατάλογο λεπτομερώς, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ε, σε, αντιπαράθεση με την Πολωνία για το benchmarking. Ε, βλέπουμε θέματα, βλέπουμε που διαπίστωσαν περισσότερε που είχαν περισσότερες δυσκολίες η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Υπήρχαν όμως λίγε λίγες περιοχές, λίγοι τομείς, όπου οι χώρες είχαν λιγότερες δυσκολίες από την Πολωνία. Πολύ λίγες όμως. Και παρά τα απορίσματα που ανέφερα προηγουμένως ότι αφορά ας πούμε, τη δημιουργία του, καλά, κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τα διαφορετικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Εδώ, σε ό,τι αφορά τα συστήματα συγχρηματοδότησης και τι διαδικασίε, οι δύο χώρες είχαν λιγότερες δυσκολίε από την Πολωνία. Και για το ρόλο και τα καθήκοντα για τα, τα, τους εθνικούς φορείς και τους περιφερειακούς ε, φορείς, το ίδιο. Παρότι τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγηση ήταν αδύναμα και οι δύο χώρες παρόλα αυτά είχαν λιγότερες δυσκολίες από την Πολωνία. Πάμε σε λίγες στατιστικές ε, σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των, της προενταξιακής χρηματοδότησης στο να δημιουργήσει μορφές ε, management ε, με βάση τα ταμεία, τα διαφορετικά ταμεία, όπως βλέπουν τα διαφορετικά ταμεία. Βλέπουμε στις 3 Νοεμβρίου ποια, ποιες από αυτές τις δομές είχαν εγκριθεί. Και βλέπουμε ότι για την ε, Βουλγαρία τίποτα δεν είχε εγκριθεί, ενώ στη Ρουμανία κάτι παραπάνω από 75% αυτών των δομών είχαν εγκριθεί. Εν συνεχεία, ε, το ποσοστό πληρωμής του Διευθυντικού Ταμείου στο τέλος του 2009 είναι ένας άλλος δείκτης που χρησιμοποίησαμε. Για τη Βουλγαρία βλέπουμε ότι είναι 9% και για τη Ρουμανία είναι 10%. Αυτά δεν είναι τα χαμηλότερα ποσοστά πληρωμών. Η Ολλανδία είχαν 7%. Μέχρι το τέλος του 2010 η κατάσταση άλλαξε λιγάκι. Η Βουλγαρία έφτασε στο 15% ποσοστό πληρωμής και η Ρουμανία μικρότερη αύξηση είχε, έφτασε στο 13%. Αξιοσημείωτο είναι ότι για τα περισσότερα κράτη-μέλη τα ποσοστά πληρωμών είχαν αυξηθεί πολύ πιο σημαντικά, πολύ περισσότερο υπήρχαν και κάποιες ιστορίες έτσι, επιτυχίας, παρά τις σημαντικές δυσκολίες και, παρά, και παρά τις ελλείψεις, η εισαγωγή προγραμμάτων και σχεδίων ως αναπτυξιακά εργαλεία θεωρείται επιτυχία, δεδομένης της αφετηρίας των δύο χωρών όταν ξεκίνησε η προενταξιακή χρηματοδότηση. Και παρότι υπήρχαν δυσκολίες στην ε, εμπλοκή διαφόρων stakeholders, μίλησα για την αρχή της εταιρικής σχέσης προηγουμένως και τις δυσκολίε που υπήρχαν. Παρ' όλα αυτά, η συμμετοχή αυτών των φορέων, αυτών των stakeholders, είχε βελτιωθεί σημαντικά ε, σε σχέση με την στιγμή κατά την οποία ξεκίνησε η χρηματοδότηση. Και παρότι υπήρχαν αδυναμίες στα συστήματα management και ελέγχου, αν συγκρίνουμε την κατάσταση πώς είχε στην αρχή η κατάσταση τελικά βελτιώθηκε σύν το χρόνο. Αξιοσημείωτο είναι επίσης η αύξηση της ε, διαφάνειας και της και η ικανότητα των ε, κεντρικών και περιφερειακών αρχών να λογοδοτούν ε, σε ό,τι αφορά τις αδυναμίες για την ε, δημιουργία τέτοιων δομών Μία δυσκολία που αντιμετωπίσαμε είναι ότι η έκθεση της Κομισιόν δεν δίνει στοιχεία ή δίνει λίγα στοιχεία για τη συνεισφορά της προενταξιακής υποστήριξης, δηλαδή για το κατά πόσο ήταν αποτελεσματική. Ως προς τον προσδιορισμό αυτών των στοιχείων. Και ανέφερα νωρίτερα ότι γενικέ προσδοκίε ω προ ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν ε, τα προενταξιακά προγράμματα και σχέδια ήταν μάλλον ουτοπικέ υπήρξε μια ασταθής και βραδία πορεία μέχρι την προσχώρηση η οποία μάλιστα άφησε πολλά κενά που έπρεπε να συμπληρωθούν ε, στην ε, περίοδο που ακολούθησε την ε, ένταξη. Η ίδια η προενταξιακή περίοδος δεν ήταν επαρκής για τη λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων και ταμείων συνοχής, δηλαδή δεν επετράπει η ανάπτυξη θεσμών τέτοιων που να μπορούν να συμμετέχουν στη διαχείριση των ορθωτικών τομείων ή ουσιαστικά να συμμετέχουν. ή δεν προσεφέρθησαν από την ε, ε, διοίκηση οι σχετικές δυνατότητες για ανάπτυξη αυτών των πόρων, ακόμα και όταν υπήρχαν οι θεσμοί. Και επίσης η Βουλγαρία και η Ρουμανία παρέμειναν εξαρτώμενες για τεχνική υποστήριξη και μετά την προσχώρησή τους από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ε, επιχείρημα που παρουσιάστηκε πλέον σε εμά ότι και άλλα κράτη-μέλη μπορεί να ερμηνεύουν όπως θέλουν τους κανόνες και τους κανονισμούς ενώ φαίνεται ότι ε, η Κομισιόν μπορούσε να τις απαλλάξει από ένα μέρος του φόρτου εργασίας. Εν όλο λοιπόν διδάγματα και συστάσεις ως εξή. Το προενταξιακό μέσο είναι καταλληλότερο ως μέσο υποστήριξης της περίοδου, στην προενταξιακή περίοδο για τη μελλοντική διαχείριση με δεδομένο ότι οι θεσμοί και οι δομές που εφαρμόζουν το πρωταξιακό μέσο τώρα θα είναι οι ίδιοι δομέ και, ε, δομές και θεσμοί που θα το εφαρμόζουν στο μέλλον, δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να δούμε τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι θεσμοί μπορούν να προχωρήσουν προς την ανάπτυξη των δυνατοτήτων που απαιτεί η διαχείριση των διευθυντικών ταμείων. Και έτσι φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να υπάρχει πιο, θα πρέπει μάλλον να υπάρχει πιο αυστηρή αξιολόγηση της ε, δυνατότητας διαχείρισης των πόρων. στην πράξη και όχι επί χάρτου όπως είναι μέχρι τώρα. Θα προτείναμε όρους και προϋποθέσεις για την ενισχυμένη διαχείριση των ταμείων στο μέλλον από τις ε, υποψηφίες χώρες κατά την στιγμή της προσχώρησης. Ε, είχαμε την εντύπωση ότι η δυνατότητες και το δυναμικό αυτών των κρατών δεν αξιοποιήθηκαν στο έπακρον από τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ίσως βέβαια να εξαρτάται και από την δυνατότητα ε, συμμετοχής στη διαδικασία αυτοκρατών. Ένα σημείο ε, ήταν το σχετικό με την προενταξιακή περίοδο και τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, να αλλάξει νοοτροπία η χώρα ε, και να μπορέσει η κοινωνία των πολιτών να υποχρεώσει την διοίκηση της, την κυβέρνηση της σε λογοδοσία. Και έτσι λοιπόν είχαμε ως θέμα την, ε, το ενδεχόμενο δημοσίευση της έξιδες αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της υποχρέωσης για λογοδοσία. Οι εκθέσεις κάλυψαν που κάλυπταν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και βέβαια ξεκίνησαν το 2004, στη μεγαλύτερη τους πλειονότητα δεν ε, διετέθησαν στο κοινό. Πράγμα το οποίο θεωρούσαμε ότι θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο μέσον και για τους πολίτες στα υποψήφια κράτη και στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να υποχρεώσουν οι πολίτες σε λογοδοσία τους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης θεωρήσαμε από, το, από την ενημέρωση των διαφορών εμπλεκομένων ε, φορέων ότι χρειαζόταν καλύτερη στάθμιση της ποιότητας με την ποσότητα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή υπήρχε γενικά η εντύπωση ότι κάποιες αδυναμίες ως προς, την, ε, ε, ως προς τις διαπιστώσεις των εκθέσεων δεν είχαν να κάνουν παρά με πιο περίπλοκες προϋποθέσεις οι οποίες οδηγούσαν στην καταγραφή ε, αρνητικού προσήμου σε μια έκθεση για ένα συγκεκριμένο τομέα. Ήταν περίπλοκες δηλαδή γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Στο παρελθόν επίσης υπήρχε η πρακτική της ε, επιλογής προσωπικού ε, που θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτά τα ποσά με ανταμοιβή μισθού υψηλότερου από τον μέσο όρο, το οποίο όμως απεδείχθη εσφαλμένο και οδήγησε σε ε, παράλογα υψηλή αμοιβή για ορισμένους ολίγους αξιωματούχους που καλούνται να διαχειριστούν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να θεωρήθηκε αυτό βραχυπρόθεσμο ως λύση, αλλά πάντως δεν ήταν βιώσιμη λύση. Και πιστεύω και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, διαπιστώνεται ότι δεν είναι πάντοτε η καλύτερη λύση αυτή. Νωρίτερα αναφέρθηκα στην δυσπιστία μεταξύ πολιτών και υπαλλήλων και τις σχετικές διαδικασίες. Και είπαμε ότι θα πρέπει οι ευρωπαϊκές αρχές να ερμηνεύουν με υπερβολικά ε, περίπλοκους κανόνες και διαδικασίες τους ε, την ομοθεσία την ευρωπαϊκή. Δηλαδή να ξεπερνούν σε περιπλοκότα το αρχικό πεδίο και το στόχο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Γιατί αυτό βέβαια περιπλέκει πολύ τα πράγματα και δεν οδηγεί στις βέλτιστες δυνατές αποφάσεις και εν τέλει μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα ειδικό καταγραφής των αποκομιστέντων διδαγμάτων που έχουμε στη θέσή μας πλέον με πληθώρα παραδειγμάτων από τις ε, δύο τελευταίες διευρύνσεις, 2004 και 2007, και που δεν έχει ληφθεί υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ευχαριστώ και εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίασή μου. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ εκ βάθους. Ε, νομίζω ότι έχουμε... Ε, τώρα ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο για να θέσει ερωτήματα. Η κυρία Ιβάνοβα. Κάποιος άλλος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την ε, εταιρεία συμβούλων που έκανε το έργο αυτό και ευχαριστούμε και τη γραμματεία η οποία έκανε τις προδιαγραφές επί τη βάση των οποίων θα πρέπει να εκπονηθεί αυτή η μελέτη. Ένας από τους κύριους στόχους μας εδώ θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα κατημέλη και οι ευρωπαϊκοί θεσμικοί οργανισμοί θα διδαχθούν από τα σφάλματα του παρελθόντος, θα ενισχύσουν τα θετικά στοιχεία και θα αποτρέψουν επανάληψη των ίδιων προβλημάτων. Με το να δούμε τα πορίσματα αυτής της μελέτης, βλέπουμε ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα για να προχωρήσουμε από τα προηγούμενα προβλήματα που υπήρχαν. Ήταν πολλές οι λήψεις και τα προβλήματα και οι τωρινέ υποψήφιε χώρε τώρα έχουν καταφέρει σε ορισμένο βαθμό να λειτουργήσουν καλύτερα. Αυτό όμω οφείλεται και από την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει επιτευχθεί με την ε, εμπειρία των ενταξιακών προγραμμάτων για τα ενεστώτα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση θα βοηθήσει και την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να, δια, να μεταλαμβαδεύσουν τις βέλτιστες πρακτικές και να αποφύγουν τα σφάλματα του παρελθόντος και εδώ βρίσκεται και η προσθέμενη αξία αυτής της μελέτης να δούμε που εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στη διαχείριση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν βελτιωθεί, που υπήρξαμε επιτυχείς, που πρέπει να δαπανίσουμε περισσότερες προσπάθειες για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην χρησιμοποίηση των προενταξιακών εργαλείων. Θέλω να σταθώ σε έξι περιοχές εν συντομία, οι οποίες αναφέρθηκαν και οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για μένα στη μελέτη αυτή. Το πρώτο πρόβλημα είναι το οποίο αναφέρθηκε ήταν αυτό της διοικητικής ικανότητας. Η ανάπτυξη της διοικητικής <clears throat> ικανότητας απαιτεί μακροχρόνια και υψηλού επίπεδου δέσμευση των πολιτικών αρχών. Είναι απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Επίτροπη να αντιμετωπίσει σωστά αυτή την δέσμευση της πολιτικής εξουσίας ή την έλλειψή της σαν γνώμονα για την πρωταξιακή αρρωγή. Η μελέτη δείχνει επίσης ότι υπήρχε έλλειψη κουλτούρας μάθησης και βελτίωσης μέσα στην διοικητική κουλτούρα. Αυτή η διοικητική εμπειρία είναι απαραίτητη όχι μόνο για τη διαχείριση των προενταξιακών κονδυλίων, αλλά με τη διαδικασία τη μαθησιακή αυτή θα προετοιμάσει καλύτερα και τις χώρες που είναι υποψήφιες για την διαχείριση των ε, διαφορετικών πόρων τα μέλη. Τρίτο σημείο, η αποτελεσματική εποπτεία των διοικητικών αρχών αυτών απαραίτητο για να υπάρξει σωστή εργασία μέσα στις ταχθήσεις, ταχθήσεις προθεσμίες. Φαίνεται όμως ότι η παρακολούθηση και η εποπτεία και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία ήταν ανεπαρκής και δεν έδωσαν σωστά και πλήρη αποτελέσματα. Ε, σε πολλές περιπτώσεις οι υποεπιτροπές κατά τομής παρακολούθησης δεν ήταν ικανοποιητικό στοιχείο και αντιμετωπίστηκαν οι εκθέσεις του σαν ένα απλό γραφειοκρατικό έγγραφο και όχι σαν πηγή ε, <clears throat> δράσης. Επομένως νομίζω ότι όπως είπαν και οι, οι συντάκτες της έκθεσης αντί να τεθούν πρόσθετες απαιτήσει αναφορών θα έπρεπε να εξασφαλίσουμε από την ότι λειτουργεί καλύτερα το σύστημα κατά τομείς εποπτείας που θα βοηθούσε και την οικειοποίηση και την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Μια άλλη σημαντική πτυχή η οποία αναφέρθηκε είναι η περιορισμοί ανθρωπίνων πόρων. Υπήρχε μεγάλο πηγενέλα προσωπικού και ήταν ένα μεγάλο ε, ένα σημαντικό συντελεστή στα προβλήματα που αντιμετωπίσαν και οι δύο χώρες σε επίπεδο διοίκησης. Μπορούν να αναφερθούν πολλοί λόγοι, καταρχήν η σχέση των αποδοχών με τον ιδιωτικό τομέα, η μετανάστευση του εργατικού δυναμικού, η έλλειψη προσόντων, η δυσκολίες στελέχωσης. Οι, λοιπόν, ε, οι μεγάλες αλλαγές στο προσωπικό εμπόδισαν την σωστή εφαρμογή. Χρειάζεται λοιπόν και παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής και καλή δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος για τα προενταξιακά κονδύλια. Υπάρχουν τώρα και σημεία επιτυχίας. Είναι λίγα αλλά είναι σημαντικά. Αφού δούμε όλα τα αρνητικά παραδείγματα είναι καλό να υπογραμμίσουμε ότι υπήρξαν και θετικά παραδείγματα, σημαντικές επιτυχίες σε προενταξιακό επίπεδο για να μπορέσουν να βοηθηθούν, να δημιουργηθούν οι δομές διαχείρισης των διαρθρωτικών πόρων <clears throat> και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, όπου ακολουθήθηκε μια συστηματική διαδικασία για να υπάρξει ανάπτυξη και μεταρρύθμιση και αυτά οδήγησαν σε αυξημένη ικανότητα σχεδιασμού, θέσπισης προτεραιότητων, διαχείρισης κτλ. Τι μάθαμε από όλα αυτά. Ότι τα προενταξιακά εργαλεία μας έδωσαν πολλά διδάγματα. Τώρα τα, οι απαιτήσει για τα προγράμματα IAP είναι καλύτερα ευθυγραμμισμένα με αυτά των διαρθρωτικών ε, ταμείων. Στην αρχή τα κονδύλια αυτά και τα προενταξιακά πλαίσια δεν αντανακλούσαν τις ανάγκες διαχείρισης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους. Κάτι ακόμα το οποίο αναφέρατε στην έκθεσή σας ήταν η υπερφόρτωση με απαιτήσει. Παραγωγής χάρη οι τριμηνιές εκθέσεις θα πρέπει να είχαν εξασφαλίσει μια ισορροπία μεταξύ ποιότητος και ποσότητος πολλές φορές οι υπηρεσίε τη Κομισιόν αντιμετωπίζουν δυσκολίε και ελλείψεις στην παράδοση εκθέσεων με το να ζητούν ακόμα περισσότερε εκθέσει κάτι το οποίο οδηγεί σε πρόσθετο γραφειοκρατικό άχθος αλλά δεν βελτιώνει την ποιότητα των εκθέσεων. Έχουμε δει ότι ακόμα και οι απαιτήσει της Κομισιόν μπορούν να δημιουργήσουν υπερβολικό φόρτο εργασία σε ορισμένε υποψήφίε, αλλά ακόμα και χώρε μέλη. Κλείνω με μια παρατήρηση δεν πρέπει να την αντιμετωπίσετε ως επίκριση, αλλά θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό λεπτομεριακότερα. Είναι το θέμα της συγκριτικής ανάλυσης μεταξύ των δύο αυτών χωρών και άλλων χωρών κατά τη διάρκεια της προεταξιακής τους διαδικασίας. Πιστεύω ότι η ανάλυση θα ήταν πολύ πιο ισχυρή αν είχαμε μια πιο λεπτομεριακή συγκριτική ανάλυση. Έχετε μια τέτοια σύγκριση στη σελίδα 33 σημειώτηση 4 2 που συγκρίνει τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία με την Πολωνία αλλά δεν είναι αρκετά λεπτομεριακό το σημείο αυτό για να δώσει επαρκείς πληροφορίες δεν είναι σαφές από πού έχουν έρθει τα πορίσματα, πώς έχουν επιλεγεί τα κριτήρια σύγκρισης εκεί που γίνεται η σύγκριση. Αναφέρεται ότι οι δύο χώρες αυτές λειτουργήσαν χειρότερα σε ένα τομέα και καλύτερα σε έναν άλλο. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε πιο πλήρη πορίσματα στα θέματα αυτά και να ακόμα σημείο την Κροατία και την Ισλανδία που είναι και αυτό τμήμα της ανάλυσης της συνδετικής για μένα δεν φάνηκε αυτό σαν σύγκριση ουσιαστικά αλλά απλώς σαν μια σύντομη ανάλυση της κατάστασης στην Ισλανδία και στην Κροατία δεν εμπεριείχε όμως τα συνδετικά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποια σύνδεση με την Βουλγαρία και την Ρουμανία που ήταν το αντικείμενο αυτή τη μελέτη. Παρ' όλα αυτά, σα ευχαριστώ πολύ για την εργασία σα και σα συγχαίρω. Ευχαριστώ κυρία Ιβάνοβα. Άλλοι δύο θα αναλάβουν το λόγο. Ο κύριος Μπαλτσίτης και μετά η κυρία Γκρέσλε. Τέλο η Κομισιόν. Κύριε Μπαλτσίτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες αυτές και επίκαιρε. Να, το να μιλάμε δηλαδή για την εμπειρία της συναδέλφου της κυρίας Ιβάνοβα, να δούμε τα, τα, τα υπέρ και τα κάτω, να δούμε τις θετικές και τις αρνητικές πτυχές. Ούτως ή άλλως αυτά τα έζησαν και η Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ε, πριν από αυτές τις χώρες έγινε μια άλλη ένταξη από πολλές χώρες που είχαν αντίστοιχα προβλήματα. Ορισμένα αναφέρθηκαν στις διαφάνειες. Πριν από κάνα δύο μήνες ή μάλλον πριν από κάνα χρόνο είχα πει και θα το ξαναπώ ξανά και ξανά ότι πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα από, από αυτή την εμπειρία. Ο συντάκτης της μελέτης είπε ότι ίσως ήταν υπερβολικά πολύ οι στόχοι που έπρεπε να υλοποιηθούν. Με σχετικά χαμηλή χρηματοδότηση. Κάθε υπουργό. προσπαθούσε να εξασφαλίσει τα περισσότερα δυνατά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν η αξιολόγηση της δουλειάς του, χωρίς να ψάχνει δηλαδή να δει πώς θα απορροφηθούν τα κονδύλια και υπό ποιες συνθήκες. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να το ξαναδούμε στο μέλλον. Δηλαδή να δούμε και τους ανθρώπινους πόρους, τους ανθρώπους που δημιουργούν τα συστήματα, τους ανθρώπους που παρακολουθούν την όλη διαδικασία θα πρέπει να, είναι, να έχουν πολλά προσόντα, να ξέρουν ξένες γλώσσες, να καταλαβαίνουν περίπλοκους δημοσιονομικούς κανονισμούς και να έχουν και πολλά πολλά άλλα προσόντα ε, τους προσλαμβάνουν οι ιδιωτικές εταιρείες, οι εμπορικές τράπεζες και, τους, και φεύγουν από τη δημόσια διοίκηση. Το πρόβλημα αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Ε, Επίσης έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ της Κομισιόν, των υπαλλήλων της Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Και αυτό αναφέρθηκε. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Νομίζω ότι οι υπάλληλοι της Κομισιόν που είναι υπεύθυνοι όχι για τη χρήση των κονδυλίων, αλλά για τα συστήματα. Δεν ενδιαφέρονται να αλλάξουν τα συστήματα. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή έτσι, και τη χρήση των κονδυλίων, την αξιοποίησή τους. Υπάρχουν ε, προβλήματα, γιατί τα ποσοστά απορρόφησης είναι πάρα πολύ χαμηλά. Και συμφωνώ με την τελευταία διαφάνεια που λέει ότι θα πρέπει να μιλήσουμε όλοι για τα διδάγματα και να απορροφήσουμε, να τα χωνέψουμε αυτά τα διδάγματα. Υπάρχουν κράτη-μέλη που είναι εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προηγούμενα κύματα ένταξης, αυτά έχουν συσσωρεύσει, αυτά τα κράτη έχουν συσσωρεύσει πείρα. Έχουν πιο αποτελεσματικά συστήματα, λιγότερο γραφειοκρατικά, λιγότερο, με λιγότερες πολιτικές παρεμβάσεις και περιπλοκές. Ε, οι πολιτικοί δεν είναι εύκολο να δημιουργήσουν νέα συστήματα και να αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Γιατί ούτω ή άλλως καθώς γίνονται εκλογέ, αλλάζουν τα πρόσωπα, έρχονται οι νέοι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τις ε, εδώ προϋποθέσεις. Νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και η διαδικασία να γίνει πολύ πιο εύκολη και για την Κομισιόν και για τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέσλα. Εγώ βρήκα πολύ σε αυτή τη μελέτη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντάκτες την, ε, της έκθεσης και τη γραμματεία που την ε, έθεσε το πλαίσιο για την έκθεση και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να μάθω κάποια Πράγματα υπάρχουν κάτι τα οποία ίσως δεν κατάλαβα πολύ καλά ή δεν πρόσεξα αρκετά στην παρουσίασή σας. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα για τη σελίδα 31. Βλέπω κάτι χρώματα. Θα ήθελα να ξέρω τι λένε αυτά τα χρώματα, τι ακριβώς σημαίνουν στη σελίδα 31 και αλλού η Πολωνία είναι ως PL, αλλού είναι ως PO. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε κάποια ενότητα στα, στις συντομογραφίες για να μπορεί κανείς να παρακολουθεί το τι γίνεται. Κάτι ακόμα θέλω να σας ρωτήσω. Και τα δύο κράτη-μέλη είχαν ιδιαίτερες δυσκολίες γιατί ήταν φτωχά κράτη-μέλη. Αυτό έχει να κάνει και κάτι με το μηχανισμό επαλήθευσης. Αυτός ο μηχανισμός έχει λειτουργήσει σωστά. Τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε. <clears throat> Ξέρω ότι μπορεί να μην ήταν ακριβώς το θέμα αυτό της εκθεσής σας και μπορεί να μην έχετε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Και τώρα το θέμα της ε, διοίκησης και της ε, εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου. Υπήρξε τρόμος και φόβος από την πλευρά της δίκης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου ή έγιναν όλα με τρόπο ικανοποιητικό. Ε, δεν ξέρω τώρα αν η έκθεσή σας μπορεί να δώσει κάποια δεδομένα, αν έγιναν όλα σωστά ή όλα λάθος ή οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ σκέφτομαι και τη δική μου χώρα που είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν <clears throat> αυτά που είπατε ισχύουν για τις νέες χώρες και όχι μόνο για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, πράγματα που γνωρίζω και από τη χώρα μου, τότε θα έχουν πραγματικά πρόβλημα. Αναφορθήκατε επίσης και στην νομική βάση ορισμένων μέτρων. Μήπως έχετε κάποια πρόταση που θέλετε να θέσετε και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει αυτά τα συστήματα. Αυτό ήταν και το επόμενο ερώτημά μου. Σας ευχαριστώ τα μάλα. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι κατάλαβα πλήρως αυτά τα οποία ζητήσατε τα ερωτήματά σας. Για τα χρώματα στο γράφημα, εμείς προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε στη σελίδα 30, όπου εξηγούμε τι ακριβώς δείχνουμε στο γράφημα. Το γκρι σημαίνει ότι δεν υπήρξε κάποιος περιορισμός ο οποίος έχει διαπιστωθεί στις τακτικές εκθέσεις της Κομισιόν και η τελική στήλη αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Το κίτρινο όταν υπάρχει κάτι που αναφέρθηκε σε μία-δύο εκθέσεις, το πορτοκαλί σε τρεις-τέσσερις και το κόκκινο σε όλες τις εκθέσεις που καλύπτουν τα χρόνια χρηματοδότησης. Τώρα, κυρία Άκερμαν, συγγνώμη σας διακόπτω, Χαίρομαι που δίνετε μια απάντηση στην κυρία Γκρέσλα. Αλλά και η Κομισιόν έχει να κάνει κάποια σχόλια. Έχουμε εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, Διεύρυνσης κτλ. Μήπως θα ήταν καλύτερα προτού δώσετε πλήρες απαντήσεις η Κομισιόν πρώτη να λάβει το λόγο. Δεν ξέρω ακριβώς ποιος θέλει να λάβει το λόγο από εσάς, εσείς. Ευχαριστώ. Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Πολιτική και μαζί με την ε, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης διαχειριζόμαστε τα κονδύλια ε, των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για την ε, Βουλγαρία και τη Ρουμανία και μας υπεύθυνοι και για το μέσο προενταξιακής ενίσχυσης. συμφωνούμε γενικά με, τις, τα συμπεράσματα της έκθεσης και με τις επικρίσεις προς τις υπηρεσίες της Κομισιόν, τις οποίες δεχόμαστε. Η έκθεση εστιάζεται κυρίως σε ένα από τα τρία μέσα τα προενταξιακά, το πρόγραμμα FAR. Υπήρχαν δύο άλλα μέσα, το ISPA που ήταν ένα μέσο που είχε σκοπό να προετοιμάσει για το Ταμείο ε, Συνοχής και το SAPARD που ήταν το μέσο ε, περιφερειακής ανάπτυξης. Προετοίμασε την περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι περιορισμένο λοιπόν να, το να απομονώσουμε το ένα από τα τρία, ενώ υπήρχαν και άλλα δύο μέσα που συνδέονταν και αυτά με, τα, με την προετοιμασία των κρατών για τα διαφορετικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Ναι, Πρόεδρε, μάθαμε από την, ε, από την κακή εμπειρία του παρελθόντος και το σημερινό προενταξιακό μέσο, το είπα, έχει πέντε συνιστώσεις. Από, τις τρι, από αυτές οι τρία και οι τέσσερα, οι τρία, οι τέσσερα και οι πέντε είναι η προετοιμασία για την φάση μετά την ένταξη. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τις ίδιες δομές, τους ίδιους κανόνες, κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα ε, σε πιο μικρή κλίμακα μετά την ένταξη ή μάλλον πριν την ένταξη σε σχέση με το τι θα συμβεί μετά την ένταξη. Σε όλη αυτή την προενταξιακή προσπάθεια θελήσαμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε τις υποψήφιες χώρες ε, να μάθουν στην πράξη. Αυτό ήταν ο στόχος. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε, να υλοποιήσουμε κάποια project, ακόμα και αν δεν ήταν τέλεια, ακόμα και αν δεν υλοποιούνταν 100%, τουλάχιστον να προχωρήσουν για να πειραματιστούν οι χώρες αυτές στην πράξη τι και να δουν τι τις περίμενε μετά την ένταξη. Δύο-τρεις παρατηρήσεις τώρα για τη Βουλγαρία και η Ρουμανία. Γιατί είμαστε υπεύθυνοι για, τώρα για τη διαχείριση ε, σημαντικών κονδυλίων που αφορούν τη Ρουμανία και την ε, Βουλγαρία. Αυτές οι δύο χώρες ε, είχαν, έλαβαν πιστώσεις γενναιόδορες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξι με 7 φορές πιο σημαντικές από αυτό που μπορούσαν να πάρουν ε, δυνάμει της προενταξιακής βοήθειας. Ακόμα και αν είχαν διοικητικό δυναμικό ύψους 1, από τη μια μέρα στην άλλη μετά την ένταξη έπρεπε να εφταπλασιάσουν το δυναμικό τους. Αυτό βέβαια δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Επίσης, η Ρουμανία και η Βουλγαρία ακόμα και σήμερα έχουν τεράστια προβλήματα διοικητικά, διοικητικού δυναμικού. Και τα και το ποσοστό απορρόφησης των ε, κονδυλίων από τα ταμεία είναι πολύ χαμηλό ακόμα και σήμερα. Επίσης αυτές οι δύο χώρες τη στιγμή της διεύρυνσης, τη στιγμή της ένταξή τους δηλαδή, ε, ήρθαν αντιμέτωπες με το κοινοτικό κεκτημένο και όλοι οι κοινοτικοί κανόνες έπρεπε από τη μια μέρα στην άλλη να εφαρμοστούν όπως οι δημόσιες αγορές, οι κρατικές ενισχύσεις, ε, το περιβαλλοντικό κεκτημένο Δηλαδή τομεί όπου υπήρχαν εκατοντάδε οδηγίε που ξαφνικά έπρεπε να τεθούν σε εφαρμογή. Όχι μόνο σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έτσι λοιπόν όλοι οι εταίροι και οι δημοτικέ αρχέ τα να συμμετάσχουν σε αυτή την υπόθεση που θα αποτελούσε μια πολύ σημαντική πρόκληση και για κάθε νέο κράτο μέλο, αλλά και δεδομένου ότι υπήρχαν πολύ περιορισμένε διοικητικέ δυνατότητε, η κατάσταση ήταν μερικέ φορέ και τραγική ακόμη. Κάτι άλλο, χαρακτηριστικό πιστεύω των δύο κρατών μελών, ήταν προβλήματα διακυβέρνησης, ορατά σε κάποιες περιπτώσεις, διακυβέρνησης ή καλής ε, διαχείρισης, όπου ε, όταν έχουμε δυνατότητες σε κεντρικό επίπεδο μπορεί να μην τις έχουμε αυτόματα σε το επίπεδο τοπικών αρχών, οι οποίες καλούνται όμως με τη σειρά τους να εφαρμόσουν κάποια σχέδια που είναι και τα δικά τους ε, σχέδια ή έργα όπως σχολεία, οδόστρωση, υποδομές κτλ. που είναι αρμοδιότητα των τοπικών αρχών ήταν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι εν λόγω χώρες και ακόμη δεν έχουν θρέψει τα πράγματα. Ακόμη και τώρα, ενώ έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την προσχώρηση. Κάποια σημεία που μπορεί να αποκλίνουμε ως προς την έκθεση. Καλύτερη διατύπωση όρων και προϋποθέσεων που θα μπορούσαμε να έχουμε ε, συνδυάσει με, την, ε, με το διοικητικό δυναμικό. Το έχουμε λάβει υπόψη στο νέο μέσον, είπα, στο νέο πρωταξιακό μέσο δηλαδή, όπου ο Ευρωπαίο νομοθέτη, δηλαδή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υιοθέτησε τον κανόνα νήσιν 3. Δηλαδή εμεί δεσμευόμαστε και αν μέσα στα τρία χρόνια δεν έχουν απορροφηθεί τα μέσα, αυτομάτω αποδεσμεύονται. Πρόκειται για κανόνα που προφανώ σχετίζεται με το διοικητικό δυναμικό. Αν κάποιο δεν έχει το δυναμικό αυτό, χάνει τα κονδύλια. Πρόκειται για ένα σαφέστατο και πολύ γερό όρο που ήδη προξενεί δυσκολίε στα υποψήφια, τα τωρινά υποψήφια κράτη, γιατί θα χάσουν κάποιου πόρου στο τέλο του έτου, όπω φαίνεται. Ένας άλλος, ε, ένα άλλο σύστημα είναι η δημοσιονομική διόρθωση. Πάλι διορθωτικό μέσον, όπου βλέπουμε ε, προβλήματα ε, σφαλμένης απορρόφησης ή προβλήματα πιστοποιητικών στοιχείων, αποδεκτικών κτλ. Α, σταματούμε ή ανακτούμε. Επίσης, εκεί όπου γίνεται λόγος για περισσότερες πληροφορίες, ότι διαρκώς η Επιτροπή λογος για περισσότερε πληροφοριες οτι διαρκώ η επιτροπη ζητει ολο και πιο πολλές πληροφορίες κτλ. Με ακούλπα. Ομολογώ, μάλλον φταίω ο ίδιο Ευθέω γι' αυτό. Πλην όμω, κύριε Πρόεδρε, όταν δεν υπάρχει μελέτη σκοπιμότητα όταν δεν υπάρχει μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον. Όταν δεν υπάρχει μελέτη κόστους και αποτελεσματικότητας ή αποτελέσματος ε, σε ένα κατεθέν σχέδιο. Ε, δεν πρέπει να τους να μας τα παρουσιάσουν και αυτά. Πρέπει να παραδεχτείτε και εσείς ότι κάποια στιγμή θα ζητούμε επιπλέον πληροφορίες όταν το σχέδιο δεν έχει ε, καταρτιστεί όπως πρέπει, όταν δεν είναι όλα τα στοιχεία πλήρη πριν από την υλοποίηση. Και κάτι άλλο. Οι ανθρώπινοι πόροι έχουν κεφαλαιόδη σημασία. Λέει δε ο συντάκτη εκθέσεω ότι δεν αποτελούν λύση οι υψηλοί μισθοί. Πλην όμως κύριε Πρόεδρε, όταν είχαμε επανειλημμένες προσπάθειε κατάρτιση και διαρκή κατάρτιση πριν από την ένταξη. Και όταν μετά την ένταξη βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανεί σε θέση μα και μόνο νέοι υποψήφοι εμφανίζονται, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα για τι πράγματα τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ξαναρχίσουμε την αρχή. Περνάνε χρόνια για να καταρτήσουμε νέο προσωπικό και μετά πάλι μπορεί να χρειαστεί να ξαναρχίσουμε από το μηδέν. Και όντω λοιπόν πιέσαμε τα κράτη-μέλη και τα υποψήφια κράτη να αυξήσουν τους μισθούς έτσι ώστε να είναι ελκυστική αυτή για το προσωπικό που θα διαχειριστεί τα σχέδια και τα κονδύλια. Έτσι στο προσωπικό αυτό να μείνει μέχρι τέλους και να έχει και τη σχετική ποιότητα που απαιτείται. Αυτά είναι, Πρόεδρε, οι βασικέ μα ε, σκέψει. Και αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, ίσω θα ήθελε και ο συνάδελφο από την Γενική Διεύθυνση για τη Διεύρυνση να πει δύο λόγια για το πρόγραμμα ΦΑΡ. Ασφαλώ, λέει ο Πρόεδρο. Κύριο Ανδρέ, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τη Γενική Διεύθυνση Διευρύνσεω την είναι πρόσδεκτη φυσικά η έκθεση. Οτιδήποτε μάθαμε μπορούμε να αποκομίσουμε είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε λοιπόν ε, μελετήσει την έκθεση και το σχέδιο. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τους συντάκτες αυτής ε, κατά τη διάρκεια της ε, εκθέσεως και ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Θα ήθελα λοιπόν να περάσω στα ε, ειδικά θέματα και να σημειώσω ότι το κεκτημένο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο ΙΠΑ, στο πρωταξιακό μέσον δηλαδή, έχει ληφθεί υπόψη σε μεγάλο βαθμό του σύνολου των διδαγμάτων ε, του παρελθόντος και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 1 βλέπουμε να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά. Προσπαθούμε λοιπόν να λάβουμε υπόψη τα διδάγματα, όπως έλεγα. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι κάνουμε τη μελέτη μας, βλέπουμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε και τους δικαιούχους και ενσωματώνουμε τα δάγματα αυτά ε, σε κάθε έγγραφό μας. Καταγράφουμε δηλαδή στην επικοινωνία μας με ονδήποτε δικαιούχο την εμπειρία που έχουμε από τον ίδιο δικαιούχο, από άλλους δικαιούχους, γενικά από τη δουλειά που έχουμε κάνει στην Γενική Διεύθυνση για τη Διεύρυνση. Και επίση. Είχαμε τελευταία και εκθέσει ειδικά για το θέμα αυτό μεταρρύθμιση, τη διοικητική μεταρρύθμιση, το οποίο είναι πολύ περίπλοκο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που υπόθηκε για του μισθού, αλλά είναι αυτό και η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε την υπόθεση των υπαλλήλων γενικά του προσωπικού που έχουμε και το συζητούμε πάντοτε με τις αρμόδιες αρχές και τις κυβερνήσεις των κρατών. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Έτερος από την Επιτροπή παρακαλώ. Όχι. Η κυρία Γκρέσλε ασφαλώς θα θέλει το λόγο. Με πολύ μεγάλη χαρά άκουσα τα όσα είπε η Γενική Διεύθυνση για τα Περιφερειακά. Έτσι ακριβώς εξηγώ και στις επισκέπτες μου τι σημαίνει να είναι κανείς μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέτοια λόγια χρησιμοποιώ και εγώ. Αλλά εγώ δεν είμαι επισκέπτης. Τα ξέρω λίγο καλύτερα τα πράγματα. Και από μέσα. Έτσι λοιπόν ρωτώ το εξή. Για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου ξέρουμε τι νομοθεσίε, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα. Ξέρουμε επίση ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία είχαν περισσότερο χρόνο του από ότι άλλα κράτη. Γιατί είχαν ξεκινήσει ήδη μαζί με τα, με τα κράτη που μπήκαν το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτώ λοιπόν γιατί ήταν τόσο πολύ μεγαλύτερα τα προβλήματα και τι μέτρα ελήφθησαν έτσι ώστε τα, τα προβλήματα αυτά να αντιμετωπιστούν ή να μετριαστούν. Και παρακαλώ να καταγραφεί στα πρακτικά ότι αναμένω ότι δηλώνω απερίφραστη αναγνώριση και ε, ανεπιφύλακτη ε, προς τις προσπάθειες των ε, εκπροσώπων εδώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προσωπικού αυτής. Αλλά θα ήθελα να μάθω συγκεκριμένα τι γίνεται, τι είδους μηχανισμός επαλήθευσης υπάρχει, πώς αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, εάν βλέπει ότι θεωρεί πως θα πρέπει και στο μέλλον στα υποψήφια κράτη, στα υποένταξη κράτη να επαναληφθεί αυτός ο μηχανισμός. Κύριο Στάση. Θέλετε να Αντιδράσετε αμέσω. Ε, Κομισιόν, ίσως καλύτερα να δώσω το λόγο στον κύριο Άκερμαν πρώτα να κάνει ένα σχόλιο. Πολύ σύντομα, γιατί σε λίγα λεφτά πρέπει να φύγω. Να αναφερθώ σε κάποια ερωτήματα για τους μηχανισμούς επαλήθευσης. Μας ζήτησαν ρητός να μην καλύψουμε αυτό το σημείο. Γι' αυτό λοιπόν η έκθεση δεν μπαίνει σε αυτό το σημείο σε αυτό το θέμα. Για τα σχόλια της Γενικής Διεύθυνσης ε, για την Περιφερειακή Πολιτική. Στην πρώτη σελίδα η έκθεση αναφέρεται όντως το κυρίως στο ΦΑΡ, αλλά όχι μόνο. Λάβαμε υπόψη τα μέλη και υπάλληλοι της ε, Επιτροπής και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι έκαναν σχόλια για τα άλλα δύο, τις άλλες δύο συνιστώσεις, το ΙΣΠΑ κτλ. Και υπάρχουν κάποιες αναφορές σε βασικά σημεία. Αλλά εστιάσαμε την προσοχή μας πιο συγκεκριμένα σε κάποιους τομείς, ούτω ώστε να εμβαθύνουμε σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς. Εμβαθύναμε λοιπόν παρά να σκιαγραφίσουμε έτσι μια χοντροειδή εικόνα. Ε, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να είχαμε μπει τόσο βαθιά αν είχαμε καλύψει και τις άλλες δύο συνιστώσεις. Τώρα, ε, για την ε, διαδικασία μάθησης, ότι μαθαίνει κανείς στην πράξη. ένα σχόλιο που το έκανα και οι υπηρεσίες της Κομισιόν, αλλά και οι stakeholders, ήταν ότι ενεπλάκει πολύ το προσωπικό της Κομισιόν στη διαχείριση των σχεδίων των project. Και έτσι οι δύο υποψήφιες χώρες μόλις ε, δεν μπόρεσαν να μάθουν στην πράξη όσο περιμέναμε. Γι' αυτό είπα λοιπόν ότι θα έπρεπε να αφήσετε μερικά project έστω να αποτύχουν. Ενώ εσείς είχατε την τάση να μην αποτύχει τίποτα. Αυτό θέλατε. για το τοπικό διοικητικό δυναμικό. Αυτό το αναφέρουμε στην έκθεση. Φυσικά δεν μπορούσαμε να πούμε σε όλες τις λεπτομέρειες την παρουσίαση. Για το ότι ζητούνταν υπερβολικά πολλές πληροφορίες. Αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο. Και αφορά κυρίως την παρακολούθηση. Ε, στην τελική περίοδο της προενταξιακής φάσης. Δεν είχε γίνει σωστά το monitoring, η παρακολούθηση. Δεν αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα. Υπήρχαν κάποιε προποθέσει, αναφέρονταν κτλ. Αλλά το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε. Τώρα, η μισθή των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό είναι άποψη των διαφόρων ενδιαφερομένων, των διαφόρων ε, stakeholders. Δεν είναι προσωπική η γνώμη αυτή. Εμείς απηχούμε στην έκθεση αυτή απόψεις ε, που μας μετέφεραν κάποιοι από τους ενδιαφερόμενους. Και ούτως ή άλλως και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της Κομισιόν επίσης κάνουν τέτοια σχόλια και ένα-δύο εκπρόσωποι των δύο ενδιαφερομένων χωρών, των δύο εν λόγω χωρών. Ότι οι μισθοί αυτοί και ότι, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και οι υψηλοί μισθοί δεν αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Εδώ υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στις βραχυπρόθεσμες ανάγκες να εξασφαλίσουμε καλή διαχείριση μεγάλων ποσών και την μακροπρόθεσμη ανάγκη να κρατήσουμε ένα επίπεδο στην δημόσια διοίκηση. Για τη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνση και τα σχόλια που έκανε η Γενική Διεύθυνση Διεύρυνση. Ε, ζητώ συγγνώμη που θεωρείτε ότι δεν είχατε την ευκαιρία να συζητήσετε μαζί μας ή να σχολιάσετε το σχέδιο της έκθεσης. Είχαμε παρόλα αυτά συναντήσεις με αρκετούς εκπροσώπους της Γενικής Διευθυνσής σας, της Γενικής Διευθυνσής Διεύρυνσης. Και εγώ προσωπικά μάλιστα ζήτησα α, να έχω κάποιες επαφές, μία συνάντηση μάλιστα, σε μία συνάντηση μου είπατε ότι όχι, δεν, δεν μπορούμε να γίνει, να γίνει αυτή. Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να έρθω σε επαφή και με άλλους ανθρώπους, αντίθετα. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο έκθεσης, το πώς κυκλοφορεί η έκθεση εκφεύγει του ελέγχου μα. Εμεί τη γράφουμε, αλλά δεν, την, δεν είναι ιδιοκτησία μας. Η διαδικασία ξεφεύγει από τα χέρια μας, το που θα κυκλοφορήσει δεν το ελέγχουμε. Τώρα, προσπάθησα να απαντήσω όσο καλύτερα μπορούσα στις ερωτήσεις. Ζητώ συγγνώμη. Α, πρέπει να φύγω τώρα γιατί έχω ένα αεροπλάνο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την συμβολή σας, για την μελέτη και φυσικά θα παραμείνουμε σε επαφή και ευχαριστούμε και για τις απαντήσεις σας προφανώς. Ίσως η Κομισιόν θα ήθελε να απαντήσει το πάρα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα της κυρίας Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα τη κυρία Γκρέσλε σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τους λόγους για τους οποίους η εφαρμογή του στα νέα κατημέλη του ευρωπαϊκού δικαίου, του ενωσιακού δικαίου είναι τόσο πολύπλοκη. Η προενταξιακή περίοδος έχει σαν στόχο να επιτρέψει στις υποψήφιες χώρες να αλλάξουν την νομοθεσία τους μέχρι ότου φτάσουν πλήρη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο. Αυτή είναι και, αυτός είναι και ο στόχος της διαδικασίας προεντάξης και το διάστημα αυτό δημιουργούμε και τα, τα σχέδιά μας. Αυτό δεν συνδέεται με συγκεκριμένε αλλαγέ βέβαια. Με το δίκαιο, παραδείγματο χάρη. Έχουμε θέματα κρατικών επιδοτήσεων, περιβαλλοντικού δικαίου, δημοσίων προμηθειών, σε όλες αυτές τι περιπτώσεις πρέπει να αλλάξει η υποψήφια χώρα σταδιακά την νομοθεσία της. Το ότι έχει εγκριθεί βέβαια μια νομοθεσία από το Κοινοβούλιο δεν σημαίνει ότι όλες οι περιφερειακές, τοπικές και εθνικέ αρχές θα εφαρμόσουν αμέσως τις αλλαγές. Εδώ βρίσκεται και το θέμα της συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο και της πλήρους εφαρμογής <clears throat> της συμμόρφωσης αυτής. Γι' αυτό έχουμε ακόμα προβλήματα ακόμα σε θέματα παραδείγματος δικαίου, ανταγων... δικαίου προμηθειών ή δικαίου περιβάλλοντος. Οι εθνικές αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για τα προγράμματα αυτά δεν ξέρουν πολύ καλά και την εθνική του νομοθεσία η οποία έτσι αλλιώς έχει μόλις αλλάξει. Ή μπορεί να προτιμούν τους παλιούς κανόνες οι οποίοι ήταν πιο ευέλικτοι και τους δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στην χρήση των κονδυλιών. Εκεί βρίσκονται τα προβλήματα. Σας ξαναλέω. Αν έχετε πλήρη διοικητική ικανότητα, μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα αυτά. Σίγουρα όταν η Ισλανδία γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα αντιμετωπίσουμε τέτοια μακροχρόνια ή δυσεπίλητα προβλήματα. Αλλά χώρες, χώρες που δεν έχουν ισχυρή διοικητική δομή έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Λιγάκι να πω και για τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι γεγονός ότι η πληρωμή πριμ και μπόνους στους διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν συνάδει με την έννοια της ίσης μεταχείρισης. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο είναι εύκολο να το εφαρμόσει κανείς σε μια δημόσια υπηρεσία. Αυτό που προσπαθούμε <clears throat> να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι αποδοχές είναι αρκετά ελκυστικές ώστε να αποτρέψουν αυτά τα άτομα που είναι στι δημόσιε υπηρεσίε και διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα να φεύγουν κάθε έξι μήνε και να πηγαίνουν κάπου αλλού. Οι συνάδελφοί μου στην Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση, και εγώ συμφωνώ με αυτό, θα χαιρόντουσαν πάρα πολύ να μπορέσουν να διαβάσουν εγκαίρω ένα σχέδιο αυτή τη έκθεση, ώστε να βρουν οποιασδήποτε λάθη ουσία. Καταλαβαίνουμε ότι ο, ο συντάξη έχει το δικαίωμα να επικρίνει την Κομισιόν. Αλλά ένα παράδειγμα εδώ έχουμε ένα πίνακα ο οποίος αφορά την πρόοδο που είναι στο τέλος του 2009 για τα διευθυντικά ταμεία σε όλα τα κράτη-μέλη. Εδώ η πραγματικότητα είναι ότι στο, το 2009 το μόνο που πληρώσαμε ήταν οι αυτόματες προκαταβολές. Αν είναι 7% μονάχα το ποσό για τις κάτω χώρες, είναι γιατί υπάρχει κατοχωρήτικος πλούτος ενώ σε χώρες όπως η Ρουμανία ήταν 10%. Αλλά καμία από τις δύο αυτές χώρες δεν εφήρμοσε κανένα πρόγραμμα. Θα πρέπει να δούμε τι καταβλήθηκε στις χώρες αυτές υπό μορφή πραγματικών επιστροφών για προγράμματα τα οποία είχαν εφαρμοστεί. Και υπολείπεται πολύ η Βουλγαρία και η Ρουμανία των άλλων χωρών σε ό,τι αφορά την ε, απορρόφηση κονδυλίων. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας έδινα το λόγο, αλλά με προλάβατε. Και απαντήσατε και το ερώτημα της κυρίας Γκρέσλε, για το οποίο σας είμαι ευγνώμων. Θα ήθελα τώρα να κλείσω αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Μόνο 40 λεπτά μας χωρίζουν από το τέλος της συνεδρίασης. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έλαβαν μέρος στη συζήτηση και ιδίως στην Κομισιόν πάμε στα σημεία 8 και 9. Η απαλλαγή απαλλαγή για την ΕΜΕΑ και το, την Αστυνομική Ακαδημία. Δεν μπορούσε να είναι εδώ ο κύριος Σταυρακάκης. Ο κύριος Γκάιερ πρότεινε να <clears throat> συνεξετάσουμε τα δύο θέματα αυτά, το 8 και το 9, και έχουμε και εκπροσώπους του, της Αστυνομικής Ακαδημίας και της ΕΜΕΑ μαζί σας. Κύριε Γκάιερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Μπαρτ. Είναι και η Γιούτα εδώ. Έχουμε όσο χρόνο θέλουμε λοιπόν για να συζητήσουμε με τους εκπροσώπους των δύο αυτών φορέων. Είναι βέβαια Τετάρτη απόγευμα. Τελευταία εβδομάδα επιτροπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματο του Γιώργου Σταυρακάκη που δεν μπόρεσε να είναι παρόν. Εγώ εξ ονόματο τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών των αντικαθιστώ για τους πολλαπλούς συναδέλφους που έχουν μείνει εδώ, πολυάριθμους συναδέλφους, για να εξηγήσω πώς κινείται η απόφασή μας, η θέση μας για την απαλλαγή. Εγώ χαιρετίζω την παρουσία του Διευθυντή της ΕΜΕΑ, που τον έχουμε ήδη συναντήσει προηγουμένως, και τον, τον αναπληρωτή Διευθυντή της ε, ΣΥΠΟΛ, ο οποίος ήταν παρόν προηγουμένως, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εδώ Ελπίζω να μην χαιρετώ τους στίχους και να είναι παρόν. Και επίσης χαιρετίζω τον κύριο Σέι από το ελεκτικό συνέδριο και θέλω να τον ευχαριστήσω εξ ονόματος του κύριου Σταυρακάκη για τη συνεργασία που επέδειξε. Και θέλω επίσης να σας πω ότι για διαφόρους λόγους σε ό,τι αφορά τη διαδικασία απαλλαγή είχαμε αποφασίσει ότι δεν μπορούσαμε ακόμα να δώσουμε την απαλλαγή για την ΕΜΕΑ και την Αστυνομική Ακαδημία και θέλαμε να έχουμε μερικές πρόσθετες πληροφορίε. Καταρχήν, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε την απαλλαγή για τους δύο αυτούς φορείς. Είναι κάπως διαφορετικοί οι λόγοι. Από ό,τι μου εξήγησε ο κύριος ε, Σταυρακάκης. Ε, μπορώ να παρουσιάσω τους λόγους αυτούς. Ξεκινώ με, το, με την υπηρεσία φαρμάκων. Έχουμε βέβαια ενδιαμέσως πάρει και άλλα έγγραφα που αναφέρονται και οι απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την ε, καθυστέρηση της απαλλαγής και απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν στη διαδικασία απαλλαγής του 2009. Από εμά υπάρχει ένα δεύτερο έγγραφο. που αναφέρει σε ένα κατάλογο ποιες προσπάθειες έχουν γίνει μετά από την αναβολή της ε, απαλλαγής. Παρ' όλα αυτά χρειαζόμαστε ακόμα κάποιες πληροφορίες για την ε, αντιμετώπιση ορισμένων διαδικασιών, ιδίως για συγκρούσεις συμφερόντων. Ο εισηγητής λοιπόν είχε ζητήσει για μια συγκεκριμένη περίπτωση που αφορούσε εμπειρογνώμονες και είχε ζητήσει να δει σε ποιο βαθμό είχε γίνει η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για να αντιμετωπιστούν ορισμένα προβλήματα προμηθειών. Για την ε, ε, ΣΥΠΟΛ υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα. Υπήρξαν και εδώ εμπρόθεσμες απαντήσεις στα ερωτήματα που υπήρχαν. Αναφέρονται οι πρόοδοι που επιτέθησαν με τη νέα διοίκηση, ότι έχουν γίνει σωστές κινήσεις. Και θέλω να αναφερθώ και στην εφαρμογή του πολιτού σχεδίου 2010-2014, το γνωρίζουμε από τον προηγούμενο χρόνο. Είναι ένα σχέδιο το οποίο δημιουργήθηκε με την επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει 12 στόχους, οι οποίοι θα πρέπει να καταμετρηθεί η επίτευξή τους με συγκεκριμένα ορόσημα. Ο εισηγητής αναφέρει ότι υπήρξαν κάποιες πρόοδοι στα θέματα αυτά και θα ήθελα και με την εντολή του εισηγητή <clears throat> να και προσωπικά να ευχαριστήσω το ελεκτικό ε, συνέδριο για τις έρευνες που έκανε σε ό,τι αφορά την υλοποίηση αυτού του πολιετούς σχεδίου. Θέλω να ευχαριστήσω και το ελεκτικό συνέδριο για τις απαντήσεις, για τις, τα σχόλια που μας έδωσε και τους εκπροσώπους των αποκεντρωμένων φορέων για τις απαντήσεις και επίσης για τη συμβολή των συναδέλφων που είναι ακόμα εδώ, την κυρία Χαου δηλαδή. Επομένως, εγώ ελπίζω ότι θα υπάρξουν και άλλες πληροφορίες μετά από το καλοκαίρι. Βρισκόμαστε λοιπόν σε καλό δρόμο για την χορήγηση της απαλλαγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας προτείνω λοιπόν να ακούσουμε τους ανθρώπους από τους ε, οργανισμούς, τον κύριο Σέντρα από την ε, ΣΕΠΟΛ και τον κύριο Οσί από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο κύριος Σρέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα θετικά σχόλια είναι πολύ σημαντικό για την υπηρεσία μας, για τον οργανισμό μας. μετά από τα σχόλια που υποβάλαμε, ή μάλλον από τις προφορίες, ε, θα ήθελα να σχολιάσω κάποιες τελευταίες εξελίξεις μετά τις επικρίσεις που έγιναν προς εμάς. Μετά την αξιολόγηση που έγιναν, λάβαμε μέτρα για να ε, βελτιώσουμε τη διαχείριση του οργανισμού. Και και υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις για την ε, διαχείριση γενικά της, ε, του οργανισμού μας. Ε, το Συμβούλιο Υπουργών σε μια πρόσφατη συνάντηση ε, ενέκρινε κάποια, κάποιες συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλάξαμε τη δομή, αλλάξαμε το, το σχήμα και κά, κάποιες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνονται με πιο περιορισμένη σύνδεση. Ε, όλες οι ομάδες εργασίας που δούλεψαν για την δομή θα τις ξαναδούμε για το θέμα του, τόπου, της έδρας της, του οργανισμού. Αυτό το θέμα το έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, θα το εξετάσουμε. Αλλά φυσικά απόφαση τελική παίρνει το Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Επίσης, στο μέλλον, ο κεντρικός ρόλος της, του οργανισμού θα πρέπει να ενισχυθεί και σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ψήφου της Κομισιόν, εμείς προτείνουμε να το δώσουμε αυτό το δικαίωμα ψήφου στην Κομισιόν. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται νέα εντολή. Υπάρχει σαφής ε, συμφωνία, ε, ούτως ώστε να σχεδιάζουμε στο μέλλον την ΣΥΠΟΛ με βάση μια ανάλυση αναγκών. Αυτά, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας να τις απαντήσω. Eh, ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος της ΕΜΕΑ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Ευχαριστώ καταρχάς που μας δίνετε την ευκαιρία για άλλη μια φορά να τοποθετηθούμε στη δικασία για την απαλλαγή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10 Μαΐου αποφάσισε να καθυστερήσει την ε, απαλλαγή, την απαλλαγή μας. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση, δεδομένου ότι δεν σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση τη Επιτροπή Ελόγου του Προπολογισμού. Έχουμε διάφορε αποφάσει λάβει, αλλαγή στρατηγική, ε, τοποθετήσει, οι οποίε έχουν ενσωματωθεί και ανακοινωθεί, κοινοποιηθεί στο Κοινοβούλιο σε ένα έγγραφο τον Ιούνιο. Χωρίς να υπησέλθω στις επιμέρους λεπτομέρειες, θα ήθελα λακωνικά να επισημάνω ορισμένα ζητήματα και κυρίως το τι τροποποιήθηκε στη δικασία για τις αναθέσεις, όπου είπε και γιατί ότι θα πρέπει να εισαγάγουμε μακροπρόθεσμη ε, μακροπρόθεσμο προγραμματισμό έχει ήδη πραγματοποιηθεί ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός δηλαδή για όλη τη διαδικασία για, για όλες τις ε, ε, αναθέσεις μας για τους ελέγχους και για την κατάρτιση του προσωπικού και επίσης ε, παληθεύονται όλες τις συμβάσεις από τη νομική μας υπηρεσία. Και η νομική υπηρεσία παρακολουθεί τις διαδικασίες του συνολό Έχουμε επίσης ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα για τις αναθέσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε το αρχαιακό σύστημα της μαρχιοθέτησης των εγγράφων μας επίσης εξυγχρονίζεται και συμπληρώνεται. Η δε προστασία του προϋπολογισμού μας από δεκιμάνσεις ισοτιμίες έχουν, έχει εξασφαλιστεί με την συντόμευση των προθεσμιών. Πρέπει να σας πω βεβαίω ότι από την εποχή από την οποία αποφασίστηκε ότι μετατρέπεται ο προπολογισμό μας σε σταθερό ευρώ, ενώ εμείς έχουμε να κάνουμε πληρωμές ύψους 80 έως 90 εκατομμυρίων ε, λιρών Βρετανικών, ε, προφανώς Προφανώ εξαρτάται η εκτέλεση του προπολογισμού σε μεγάλο βαθμό από τι ε, νομισματικέ ισοτιμίε. Και θα ήθελα να επισημάνω και για τους συναδέλφους από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι έχουμε κάνει σημαντικές ε, προσπάθειες για να, τροπο, για αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι, μεταφορ, οι μεταφορές κονδυλίων, αλλά δεν είναι δυνατόν πάντοτε να αποφύγουμε σχετικά μεγάλα ποσά ε, μεταφορών. Αυτό θα ήθελα να το συζητήσω διμερώς με τους αδέλφους από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ένα θέμα στο οποίο θα ήθελα να επισέλθω επιπλέον και που αποτελεί ίσω και το κύριο σημείο επίκριση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων. Η συγκρούση συμφερόντων πάντα, και η πρόληψή του είναι πάντα ένα περίπλοκο ζήτημα δεν μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζονται μέσα από ένα σταθερό πακέτο μέτρων που μπορεί να εισαχθεί κάπου, γιατί πάντα οι συνθήκε αλλάζουν. Η υπηρεσία μα λοιπόν χρόνια τώρα προσπαθεί και έχουμε ένα σύστημα για την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων ε, να βελτιώσουμε και τα, τα ποσοστά μας ε, στα φαινόμενα συγκρούσεων συμφερόντων σε επίπεδο προσωπικό ή σε επίπεδο ε, θέσεως. Αυτό λοιπόν το καταφέραμε και πέρσι και φέτος σε συνεργασία και με την Perflorex και το θέμα της συγκρούσεως προσωπικών συμφερόντων βλέπουμε ότι παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια 4-6-9, 6 διαρκως βελτίωση και ακόμη και τώρα καταγράφεται αυτή η θετική τάση. έχουμε τις δύο αρχές της, ε, του διαχωρισμού, segregation και του ε, ενώπιος ενωπίων. Έχουμε το σύστημα του peer review, τη επαλήτευση από τους ομοτήμους. Έχουμε στην τελική φάση μιας ε, απόφασης τον αποκλεισμό του αρμόδιου που έχει παρακολουθήσει την υπόθεση αυτή από τελική απόφαση και προσπαθούμε, καθώς έχουμε τεσσάρων ειδών προσωπικό, γιατί έχουμε προσωπικό μέσα στην υπηρεσία, το επιστημονικό προσωπικό από το δίκτυο, που απαρτίζει ουσιαστικά τις επιστημονικές μας επιτροπές, τους εμπειρογνώμονες που εργάζονται σε επιτροπές, το διοικητικό μας συμβούλιο, Τρίτον και τέταρτον, μια ευρύτατη ομάδα επιστημονικών ε, πραγματογνωμών που δεν συναντούμε όμω στην πραγματικότητα ποτέ, γιατί αυτοί βρίσκονται καθένα στο κράτο μέλο το οποίο διαβιώνει και επεξεργάζεται θέματα που έχουν να κάνουν με τι ε, σχέσει μα με τι εθνικέ αρχέ. Αυτέ λοιπόν τέσσερις τέσσερι ομάδε προσώπων προσπαθούμε να ε, στεγανοποιηθούν από οποιαδήποτε δυνατή ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, στο βαθμό που μπορούμε φυσικά. Έτσι κοιτάμε να μην έχει κανείς τα τελευταία χρόνια ε, επαμοιβή λάβει καθήκοντα από τον χώρο των βιομηχανικών, της φαρμακοβιομηχανίας δηλαδή. Ε, κοιτάμε επίσης να μην έχουν μετοχές από φαρμακοβιομηχανία. Μάλιστα ορισμένοι υποχρεούνται να πουλήσουν τις σχετικές μετοχές. Υπάρχει ένα μητρό των εκπροσώπων του προσωπικού και όλων των εμπειρογνωμόνων που συνεργάζονται με την υπηρεσία όπου καταγράφεται προσωπική δήλωση απουσίας, στο λόγο της τιμής, απουσίας τέτοια σύγκρουση συμφερόντων που καταγράφεται ηλεκτρονικά και από 1η Σεπτεμβρίου εφέτος δημοσιεύεται και όλας. Και έτσι μπορεί ο καθένας να επαληθεύσει τη σχετική δήλωση. Και έτσι, επίση, για να καλύψουμε όλη αυτή τη μεγάλη και γκρίζα ζώνη ε, πραγματογνωμόνων που εργάζονται για μα, αλλά δεν, τους, δεν έρχονται ποτέ στην υπηρεσία, γιατί είναι πυρογνώμονε ή πραγματογνώμονε που συνεργάζονται με τα κράτη-μέλη περισσότερα. Για να μπορούμε να του καλύψουμε λοιπόν και αυτού, έχουμε ένα μνημόνιο συνεννόηση με τις υπηρεσίες αδειοδότησης ναι, σε όλη την Ευρώπη. Ένα μνημόνιο ε, συνεννόησης λοιπόν, το οποίο ορίζει πολύ αυστηρούς κανόνες και κυρίες και κύριοι πρέπει να σας πω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο το να καταφέρουμε με 27 διαφορετικά κράτη-μέλη και 49 διαφορετικές υπηρεσίες να καταλήξουμε σε όρους και κανόνες που θα ήταν αναγνωρισμένοι από όλους κατά τον ίδιο τρόπο. Γιατί είναι διαφορετική και η αντίληψη του τι σημαίνει σύγκρουση συμφερόντων ανακράτως της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν χρειάστηκε 49 διαφορετικά μνημόνια συνεννόησης να υπογράψουμε τις αντίστοιχε υπηρεσίες. Έχουμε λοιπόν ένα ρωμαλαίο σύστημα, ένα σύστημα το οποίο ισχύει για όλη την Ευρώπη και για τη διαδικασία διοδότησης φαρμάκων. Αυτή ήταν και η καλή είδηση που είχα να σας δώσω. Η λιγότερο καλή είδηση ήταν αυτή που έχει να κάνει με την απώλεια των εμπειρογνωμόνων. Γιατί είναι τόσο ρωμαλαίο αυτό το σύστημα που τελικά αντιβαίνει στους όρους λειτουργίας, πρακτικής ε, ε, ανάπτυξης και ε, επιστημονικής εξέλιξης στα κράτη-μέλη. γιατί μην ξεχνάμε ότι γενικά στα κράτη-μέλη, γενικά στον κόσμο, συνεργάζεται η επιστήμη με την οικονομία, με το βιομηχανικό κλάδο. Εμείς ε, τους έχουμε υποχρεώσει να αποκοπούν από αυτόν και άρα υποφέρει ο επιστημονικός κλάδος στη δική μας περίπτωση. Το επισημαίνω αυτό σε ένα πρόβλημα, χωρίς να υπενήσουμε ότι θα πρέπει να υποβαθμιστούν οι ε, προδιαγραφές μας, αλλά είναι ένα πρόβλημα προς το αποτέλεσμα στη δουλειά μας. Και για να συνοψίσω, θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια μέχρι σήμερα, ώστε να ανταποκριθούμε στις επικρίσεις που έχουμε ακούσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δώσουμε ικανοποίηση στα σημεία και τις παρατηρήσεις του και γι' αυτό σας παρακαλώ εν κατακλείδη να μας χορηγήσετε την απαλλαγή. Ευχαριστώ. Eh, ευχαριστώ. Έχουμε αναβάλει την ε, απαλλαγή, ούτω ώστε να πάρουμε και άλλες πληροφορίες. Νομίζω ότι είναι καλή η διαδικασία. Πάντως ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες και από τις δύο υπηρεσίε και από τους δύο οργανισμούς, την Αστυνομική Ακαδημία και τον Οργανισμό Φαρμάκων. Έχουμε προχωρήσει στην αξιολόγηση και τώρα δίνω το λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά εμφανίζομαι εδώ και εκπροσωπώ το ε, Ελεκτικό Συνέδριο για την Απαλλαγή των δύο οργανισμών, για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Ε, μας ζητήσατε να εξετάσουμε την εφαρμογή του πολιετού σχεδίου της αστυνομίας. Εμείς ε, κάναμε το Μάιο αυτή τη δουλειά και μεγάλη χαρά σας παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα των εργασιών τον Ιούνιο, ούτως ώστε ε, να είμαστε εμπρόθεσμοι για αυτή την ακρόαση. Η έκθεση, Πρόεδρε, όπως ε, τονίστηκε, είναι γενικά θετική, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της, ε, της Αστυνομικής Ακαδημίας και συμφωνώ με τον συντάκτη της έκθεσης. Η νέα διοίκηση της ΥΠΟΛ έκανε σημαντική πρόοδο γιατί έχει προωθήσει την κουλτούρα του ελέγχου στην, στον οργανισμό. Φυσικά η λιδία αλήθως θα είναι η δημοσίευση τον ε, λογαριασμό τον Νοέμβριο για το 2010. Και δεν μπορώ να ζητήσω να αποκαλυφθούν τα αποτέλεσματα αυτού του ελέγχου εδώ στην Επιτροπή. Πιστεύω όμως ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ε, δικαιούται να είναι περήφανη για τη δουλειά της, για την επαγρύπνησή της και για τον έλεγχο που ασκεί στην ε, αστυνομική, στην αστυνομική Ακαδημία τα τελευταία χρόνια. Ελπίζω τελευταία φορά να έχουμε να κάνουμε δυσκολίε από πλευρά ΣΥΠΟΛ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, από πλευρά Ελεκτικού Συνεδρίου χαιρετίζουμε τι αλλαγέ στη διαδικασία προμηθειών που έχει ξεκινήσει ο Οργανισμό Φαρμάκων. Ε, στον ετήσιο έλεγχο όμως 2009 το είχαμε αναφέρει αυτό. Ήταν το σημαντικότερο σχόλιο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους, τον κύριο Γκάι, τον κύριο Σταυρακάκη και αν υπάρχουν οποιασδήποτε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας να τις απαντήσω. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακαβέη θέλει το λόγο. Δύο ευρωβουλευτές ζητούν τον λόγο. Κύριε Μακαβέη. Ευχαριστώ. Ε, έχω και σχόλια και ερωτήσεις. Ε, προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Όταν αναβάλαμε την απαλλαγή, ζητήσαμε συγκεκριμένες πληροφορίες και συγκεκριμένα πράγματα να κάνει ο οργανισμός. Το πρώτο αφορά την παράγραφο 35. Παραθέτω, περιμένω το διοικητικό, περιμένει το Διοικητικό Συμβούλιο να υιοθετήσει γρήγορα ένα σχέδιο δράση για να καλύψει τα προβλήματα στη διαδικασία προμηθειών μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2011. Επαναλαμβάνω, ένα σχέδιο δράσης για να καλυφθούν οι ελλείψεις της διαδικασίας προμηθειών. Αυτό που έλαβε το Κοινοβούλιο ως απάντηση δεν είναι ένα σχέδιο δράσης όμως είναι μόνο ένας κατάλογος με το σχέδιο για τις προμήθειες, με συμβάσεις όπου, που σκοπεύει να συνάψει ο οργανισμός. Δεν λέει τίποτα για το πώς θα καλύψει τα κενά της διαδικασίας των προμηθειών. Φυσικά, θα έπρεπε το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει αθετήσει και αυτό το σχέδιο δράσης. Κάτι που δεν έχει γίνει. Δεύτερο θέμα. Στην παράγραφο 31. Στο τέλος της παραγράφου λέμε. Ζητάμε από τον οργανισμό να μας δώσει την έκθεση του εσωτερικού ελέγχου από το 2007 και μετά μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή για το 2007, 2008, 2009 και 2010. Δεν λάβαμε την έκθεση. Λάβαμε μόνο ένα κατάλογο πάλι με συστάσεις ως απάντηση του οργανισμού στην έκθεση. Το θέμα με τις δημόσιες προμήθειες και αυτό το θέμα που σας αναφέρω ε, για τον εσωτερικό έλεγχο, αυτά δεν έχουν καλυφθεί. Στην παράγραφο 26, για το θέμα της σύγκρουση συμφερόντων. Μα... Αυτή η νέα πολιτική και οι νέοι κανόνες θέλουμε να μάθουμε πώς εφαρμόζονται. Επίσης, ζητάμε ένα πλήρες αρχείο για το πώ έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σύν το χρόνο. Δεν μα εστάλει τίποτα όμως προς απάντηση. Μας έστειλαν ένα αντίγραφο μιας επιστολής που έστειλε ο οργανισμός στα κράτη-μέλη, που εξηγεί στα κράτη-μέλη τη νέα διακασία που έχει υιοθετήσει για τη σύγκρουση διφερόντων. Δηλαδή ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών, όπω λέει, να επαληθεύσουν αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για τους εμπειρογνώμονες. Καμία απάντηση δηλαδή προς το Κοινοβούλιο. Μία δυσέλιδη επιστολή μας έστειλε ο οργανισμός με σε 27 αντίγραφα. Τέταρτο θέμα. Παράγραφος 23. Θέλουμε να... Είχαμε ζητήσει να ενημερωθούμε αν οι εμπειρογνώμονες και το προσωπικό ελέγχονται για την ανεξαρτησία του και πώς ε, ε, παληθεύουμε ποια είναι τα συμφέροντά τους κτλ. Δεν μας ενημέρωσαν για αυτό το θέμα. Για το πώς δηλαδή οι εμπειρογνώμονες και το προσωπικό ελέγχονται για να δούμε κατά πόσο ανεξάρτητοι ή όχι ούτε μία απάντηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μακοβέη. Νομίζω, κύριε Πότ, δεν έχετε πείσει ακόμα την κυρία Μακοβέη. Θα σας δώσω φυσικά την ευκαιρία να απαντήσετε, αλλά προηγουμένως ο κύριος Φιέλνερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω πόσες φορές έχω έρθει για να συζητήσουμε για τις υπηρεσίες κυρίως για τη ΣΕΠΟΛ, την Αστυνομική Ακαδημία, αλλά μόνο και μόνο να σκεφτούμε το χρόνο που έχουμε δαπανίσει. εφτάνει μια πια, αφήστε μας να πάρουμε μια ανάσα. Και κύριος, από το σχέση με το δικαστήριο. Αν κατάλαβα καλά αυτά που μας είπατε, μπράβο, συγχαρητήρια, καλά τα καταφέρατε ή με τι άλλο έχετε μπει στον σωστό δρόμο. Και μετά έχουμε την υπηρεσία φαρμάκων. Με κάθε σεβασμό προ την κυρία Μακοβέη. θα πρέπει αυτά που είπε να τα συζητήσουμε μάλλον στην ομάδα εργασία μα, στο ΕΛΚ. Εγώ έχω διαφοροποιηθεί στην ψηφοφορία και έχω και διαφορετική έποψη για τα πράγματα αυτά. Έχω ασχοληθεί με τις υπηρεσίες, ίσως περισσότερο χρόνο από ό,τι άλλοι συνάδελφοι, και ω μέλο και τη επιτροπή περιβάλλοντο. Αν κοιτάξουμε ορισμένα πράγματα, θα μπορούσα να πω ότι αν κοιτάξουμε ορισμένα από τα πράγματα του ψηφίσματος, ε, πολλά τα έχουμε συστήσει εμείς στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, τα έχουμε εξετάσει, τα παρακολουθήσαμε και τα παρακολουθούμε και μάλιστα καταλήξαμε και σε διαφορετικά συμπεράσματα. Χωρί τώρα να θέλω να επισέλθω σε όλη την υπόθεση και την ιστορία περί ε, διαμεσολαβητή, που υποτιθέτω ότι έπρεπε να συζητηθεί εδώ μέσα στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, τι σχέση έχει, εν περιπτώσει. Για μένα μου φαίνεται λίγο περί τη εδώ και, εν περιπτώσει, δεν αφορούσε και το φετινό έτο, τη φετινή απαλλαγή. Ε, εν πάση περιπτώσει όμως κάπου διαμέσως είμαστε μεταξύ διαμεσολαβητή και συγκρούσου συμφερόντων Ως προς την της τη και κυρίω το θέμα των δημόσιων προμηθειών έχει μεγαλύτερη ε, σχέση με τις αρμοδιότητες της ε, Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού πάνω απ' όλα. Ωστόσο, από όσα ακούσαμε και από όσα γνωρίζω και εγώ, ξέρω ότι υπήρξαν προβλήματα. Αλλά αν συγκρίνουμε τη γενικότερη εικόνα των υπηρεσιών, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος όντω για αναβολή της απαλλαγής. Και δεν νομίζω ότι θα δώσει και καμιά ουσιαστική ε, επίπτωση αυτή η αναβολή. Για μένα στο σημείο 23, Φερρυπίνου όπου ζητούμε ανεξαρτησία πραγματογνωμών και προσωπικού που θα ασχολείται με την συγκεκριμένη ουσία φαρμακευτική ε, φαρμακευτικό παρασκεύασμα κτλ. Νομίζω ότι για τη δουλειά που κάνει η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού δεν έχει θέση αυτή η διαπίστωση, η παρατήρηση. Και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον που πιστεύω ότι θα ακούσουμε και κάποια άλλα σχόλια από την υπηρεσία την ίδια. Την αναφορά δηλαδή στον παλαιό εκείνο διευθυντή ο οποίος πέρασε στον ιδιωτικό τομέα. Θα έλεγα ότι είναι μάλλον όχι πολύ κομψό και ε, σωστό. Αλλά αυτό σημαίνει ότι φταίτε εσείς. Και δεν βλέπω και πουθενά στον κανονισμό τίποτε που να ε, απαγορεύει ανάληψη δραστηριότητων στο ιδιωτικό τομέα μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία. Άλλωστε, αν ήταν κάτι τέτοιο δυνατό, θα ήθελα να το δω και για το Κοινοβούλιο. Για του πρώην Ευρωβουλευτέ δηλαδή. Πάντω, ήθελα να μου πείτε τι ε, σκέψει για την υπόθεση αυτή. Τι, Πώ βλέπετε τα πράγματα. Και κάτι άλλο για το σύγκρουση συμφερόντων. Που το θεωρώ επίση σημαντικό. Για ε, να το συζητήσουμε. Και βέβαια, για λόγου, περιβαλλοντικού, θέλω να έχετε τον καλύτερο δυνατό πραγματογνώμα, του καλύτερου επιστήμονε. Άρα το να αναστήσετε κάποιον που δεν θα έχει ποτέ εργαστεί στον χώρο τη φαρμακοβιομηχανίας και θα έχει και επαρκή και ανώτατε, μάλλον γνώσει στην υπόθεση αυτή μου φαίνεται μάλλον ουτοπικό. Γιατί όπω είπατε και εσεί, εγώ δεν θέλω τελικά να καταλήξουμε να έχουμε εμπειρογνωμόνε δεύτερη κατηγορία, γιατί εσεί αποφασίζετε ότι αποκλείεται από την πρόσληψη τέτοιου είδου εμπειρογνωμόνων που έχουν εμπειρία από το χώρο τη φαρμακοβιομηχανίας. Ερωτώ λοιπόν αντίστροφα από την άλλη πλευρά, εσά σα μεταθέτω το ερώτημα, πώ μπορείτε με την ανθεωρημένη αυτή δήλωση ε, συγκρούσεως, περί συγκρούσεως συμφερόντων, ε, πώς μπορείτε να εγγυηθείτε ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Γιατί εμεί, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος θέλουμε και ασφαλή και καλά φάρμακα να εξασφαλίσουμε πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπουμε τη δημοκρατία εν τη δράση. Πολλά μέλη δεν είναι παρόντα, λίγα είναι παρόντα, παρόλα αυτά έχουμε διαφορές απόψεων. Και πότε ίσως μπορείτε να απαντήσετε και μετά μπορούμε να δώσουμε και πάλι το λόγο στον κύριο Γκάιερ για να κλείσει εξ ονόματος του κύριου Σταυρακάκη πάντα. Νομίζω ότι για τη ΣΥΠΟΛ δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έχετε το λόγο κύριε Σεώρη. Ναι, πράγματι θεωρήσαμε ότι οι απαντήσεις στα διάφορα κεφάλαια για την, τις εκθέσεις σας θα σας ικανοποιούσαν, ιδίως σε ό,τι αφορά τα παρατήματα. Λαμβάνω όμως υπόψη τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν τα ειδικά θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα έχει δημιουργήσει μια ομάδα μαζί με τους εκπροσώπους της Κομισιόν ώστε να επανεξετάσει τις διαδικασίες προμηθειών μας, τις τροποποιημένες διαδικασίες προμηθειών. Όλα αυτά δεν είχαν γίνει μέχρι τον Ιούνιο, γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε το Μάρτιο το δρομολογήσαμε το θέμα αυτό και αποφασίστηκε στις αρχές Ιουνίου στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέσσερις φορές το χρόνο της συνεδρία του Διοικητικό Συμβουλίου χρειάστηκε αυτός ο χρόνος για να οργανωθούν τα πράγματα, αλλά θα εφαρμοστεί πια αυτή η διάταξη. Τώρα για τις ε, συστάσεις ΓΙΑΣ. Θεωρούσαμε ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου έχουν αρκετό αναγνωστικό υλικό σε σχέση με την έκθεση ΕΜΕΑ από το 2007-2008-2009 και γι' αυτό εμείς σας δώσαμε ουσιαστικά μόνο ε, ένα επίτομο έγγραφο σύνοψης αυτών τα οποία είχαν γίνει σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων για τις συγκρούσεις συμφερόντων. Κάναμε μία, ένα αγώνα που ήταν πολύ δύσκολος έχουμε από την αρχή της ύπαρξης αυτού του φορέα ένα κανόνα δεοντολογίας για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων. Στην αρχή ήταν ουσιαστικά μονάχα μια δήλωση από την πλευρά των ενδιαφερομένων. Και σήμερα ακόμα δεν έχουμε κάποια αστυνομική ή εισαγγελική διαδικασία. Βασιζόμαστε στις δηλώσεις των εμπειρογνωμών μας και τους εμπιστευόμαστε. Πρέπει να τους εμπιστευόμαστε. Και αυτό συμβαίνει με όλους αυτούς οι οποίοι αντιμετώπισαν τον Ben Fluorex στην ΕΜΕΑ, στην υπηρεσία μας. Μέχρι το 2010 το Ben Fluorex δεν ήταν σημαντικό θέμα της υπηρεσίας μας, αλλά αυτό το έχουμε συζητήσει και σε ένα άλλο πλαίσιο, γιατί βασικά ήταν ένα γαλλικό προϊόν. Για να απαντήσω στο τελευταίο ερώτημα και να κλείσω είναι πρόβλημα να έχουμε ανθρώπους υψηλού επίπεδου που να είναι εμπειρογνώμονες και επιστήμονες. Τώρα έχουμε περιορίσει πάρα πολύ την εμπειρογνωμοσύνη μας. Πρέπει να βασιζόμαστε σε εθνικούς υπαλλήλου που είναι υπεύθυνοι στα θέματα αυτά σε εθνικό επίπεδο, γιατί έχουν μια, ένα ιστορικό εργασία σε δημόσιες υπηρεσίες. Γι' αυτό δεν είναι τόσο επιρρεπής σε συνεργασία με τις φαρμακευτικές εταιρείες και ούτε είναι τα άτομα αυτά τα οποία δουλεύουν στα πανεπιστήμια και τους ζητείτε να καταφέρουν κάποια χρηματοδότηση από τη βιομηχανία. Παρ' όλα αυτά είναι ενήμεροι για τα αποτελέσματα της βιομηχανικής έρευνας. Παίρνουμε λοιπόν ανθρώπους από τον ακαδημαϊκό χώρο όπου μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι επιστήμονες στον ιατρικό και φαρμακευτικό τομέα δεν είναι αυτή τη στιγμή ή τουλάχιστον πρόσφατα εργαζόμενοι στην φαρμακοβιομηχανία. Όπως όμως είπα και προηγουμένως, αυτή η ομάδα από την οποία μπορούμε να επιλέγουμε ε, εμπειρογνώμονες γίνεται όλο και πιο μικρή όσο, και, όσο πιο σφιχτά γίνονται τα μέτρα τα οποία εφαρμόζουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάιερ θα πάρει το λόγο και θα εκπροσωπήσει τον κύριο Σταυρακάκη για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ. Και από αυτά που ακούσαμε στο παρελθόν από το ελεγκτικό συνέδριο, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η δουλειά της Επιτροπής Ελέγχου του Υπολογισμού και για την ε, ΣΥΠΟΛ και βέβαια η δουλειά του Ελεγκτικού Συνεδρίου μας βοηθάει ιδιαίτερα. Άκουσα τις παρατηρήσεις του Λεμπτικού Συνεδρίου και από τα όσα έχω δει από τον κύριο Σταυρακάκη και από τις θέσεις του μπορώ να απονομίζω χωρίς ε, να απατώμε ότι ε, βρισκόμαστε στον ίδιο δρόμο. Στα δε μνημόνια συνεννόησης ως προς το ζήτημα των ε, συγκρούσεων συμφερόντων και τη συνεννόηση στην οποία προέβηται με 49 διαφορετικέ υπηρεσίε των κρατών μελών δεν μπορεί να μας ε, είναι χρήσιμο να περιορίσουμε τόσο πολύ το πεδίο των εργασιών της ΕΜΕΑ και συμφωνώ σε αυτό ε, Φιώνα μαζί σου ότι ε, δεν θα πρέπει να περιοριστεί το πεδίο, κύριε Φιέλνερ μάλλον, δεν μπορούμε να περιορίσουμε το πεδίο εργασιών και τις δυνατότητες επιλογής της ε, υπηρεσίας φαρμάκων ε, τόσο ώστε να μην μπορεί να βρει τελικά κάποιον ε, καλό ειδικό επιστήμονα, εμπειρογνώμονα για να κάνει τη δουλειά του όπως θέλει, όπως πρέπει. Δεν μπορεί αυτό να προς το συμφέρον ούτε του ελέγχου του προϋπολογισμού, ούτε και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, ούτε και των υπηρεσιών μας. Θα ήθελα πάντως η κυρία Μακοβέη, ο σκιώδης συγγήτρια, να καταγράψει, να σημειώσει και εκείνη και να αναγνωρίσει τις πρόοδους που έχουν επιτευχθεί στην υπόθεση αυτή. Αν λοιπόν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι οι αδυναμίες που έχουμε εμείς εντοπίσει μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση κάποιων από τα προβλήματα και μας είπε και ο κ. Διευθυντής ότι συν το χρόνο τα πράγματα βελτιώνονται, περιορίζονται τα προβλήματα. Και νομίζω ότι αν μπορέσει να συμφωνήσει η κυρία Μακοβέη, νομίζω ότι καταλήγουμε στο συμπέρασμα, όπως ο κύριος Σταυρακάκης, ότι πρέπει να έχουμε έναν ορίζοντα λογικό που θα μας επιτρέψει να δούμε την επίλυση και τη μετώπιση όλων των προβλημάτων, χωρίς όμως να ε, μπορούμε να πούμε ότι λυθήκαν όλα τώρα. Αλλά πάνω απ' όλα χωρίς να μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν είδαμε να αντιμετωπίσετε και κανένα πρόβλημα ή ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό θα ήταν λάθος. Βεβαίω και πρέπει να επισημαίνουμε τα προβλήματα, αλλά ο στόχο μα θα πρέπει να είναι επισημένοντά τα να θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε κατά τρόπο ουσιαστικό. Ευχαριστώ. Θα ολοκληρώσω. Θα ολοκληρώσουμε εδώ. Ευχαριστώ όλου όσου συμμετείχαν στη συζήτηση. Ευχαριστώ το Ελληνικό Συνέδριο, του εκπροσώπου τη Αστυνομική Ακαδημία και του Οργανισμού Φαρμάκων. Έχουμε και ένα σημείο στα διάφορα. Θέλω να σας πω κάτι πριν. Για την έκθεση Σταυρακάκη, μας υποσχέθηκε ο κ. Σταυρακάκη ότι αρχές Αυγούστου θα μα στείλει το κείμενό του. Και θα έχουμε μετά ένα μήνα ε, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου το μεσημέρι για τις τροπολογίες. 22 ψηφίζουμε στην Κοκομπή και στην Ολομέλεια ε, του Οκτωβρίου ψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι κάνει κρύο τη αρκούδα αυτή την αίθουσα εγώ είμαι ήδη κρυωμένη και υποφέραδο. Προσπαθώ να επιβιώσω. Μήπω θα μπορούσαμε αύριο να ανάψουμε κανένα μαγκάλι, τουλάχιστον να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία για να υπάρχει σωστή θερμοκρασία. Υπάρχουν άτομα τα οποία πραγματικά έχουν πρόβλημα. Ευχαριστώ. Εγώ αλλιώ δεν θα έρθω αύριο. Ευχαριστώ. Υποψιάζομαι, κυρία Γκρέσλερ, ότι θα γίνετε πολύ δημοφιλείς με αυτά που είπατε.